ζωή σε αυτού Bien, chers collègues, en dépit Αγαπητοί συνάδελφοι, παρά την πολύ μικρή προσέλευση θα αρχίσουμε. Είναι απογοητευτικό αυτό, δεν το λέω για να σας απογοητεύσω, αλλά είναι και ιστορική μέρα σήμερα για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη, γιατί σήμερα τίθεται ενισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας Επομένως είναι πολύ κατάλληλος χρόνος να μιλήσουμε για την πολιτική ασφαλείας και άμυνας. Και πρέπει να αποτίσω μεν φόρο τιμής στον Χαβιέρ Σολάνα που εδώ και δέκα χρόνια με πολύ θάρρος και μεγάλη αίσθηση ευθύνης φρόντισε για την παρουσία της Ευρώπης διεθνώς και εξετέλεσε 22 διεθνείς αποστολές πολύ επιτυχής όπως κάτι που συνήθως ξεχνάμε το άτσε. Α, ευχαριστώ συνάδελφοι. Από με αμεφόρο τιμή στο Χαβιέρ Σολάνα. Ελάτε να ακούσετε. Η δράση του ήταν καθοριστική στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας όπου έγινε μια φυσικών διαστάσεων δοκιμή θα έλεγα προληπτικής διπλωματίας και έτσι η χώρα αυτή των Βαλκανίων δεν γνώρισε την τραγική τύχη που είχαν άλλες γειτονικές και αυτό οφείλεται πολύ στη δράση του Χαβιέρ Σολάνα. Νομίζω λοιπόν ότι καλό είναι να τον ευχαριστήσουμε σήμερα. Σήμερα θα μας μιλήσει η κυρία Κλαβδία Γαλλία Αρνού, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια για τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού, την οποία συγχαίρω επίσης γιατί μόλις πήρε αυτή τη θέση την Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού CMPD στα αγγλικά. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε μαζί να συζητήσουμε για τη διαδικασία που οδήγησε στην δημιουργία του οργανισμού αυτού που είναι ζωτικός για το στρατιωτικό συντονισμό και ξέρω ότι ενδιαφέρει πολλά μέλη της υποεπιτροπής μας. Θα σας ακούσουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι η εμπειρία σας θα μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να καταλάβουμε ορισμένες επιχειρήσεις που έχουν ήδη αναλυθεί όπως η Σομαλία που μας ενδιαφέρει επίσης πολύ. Επειδή έχουμε καθυστερήσει, σας δίνω αμέσως το λόγο, αλλιώς θα μιλούσα κι άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πράγματι ιδιαίτερα σημαντική η σημερινή μέρα που τίθεται ενισχύει η καινούργια συνθήκη. Εχθές ο Χαβιέρ Σολάνα ήρθε στο κτίριό μας για να επισκεφθεί το κέντρο που διευθύνω Διεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Σχεδιασμού. Τα γαλλικά σε PSS, στα αγγλικά CNPD. Λοιπόν, για να μας αποχαιρετήσει και να λήξει έτσι επίσημα η περιπέτεια αυτή την οποία από κοινού είχαμε αναλάβει. Και μας ζήτησε με μεγάλη συγκίνηση να συνεχίσουμε το έργο μας με τον ίδιο ενθουσιασμό τώρα που διαθέτουμε και περισσότερα μέσα και υπάρχει και μεγαλύτερη συνοχή στη δράση, θα υπάρχει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αφού μίλησα για συνοχή λοιπόν πρέπει να αναφέρω και το θέμα της δημιουργίας αυτής της νέας διαχείρισης της οποίας ανέλαβα τη διεύθυνση την CMPD στα αγγλικά όπως προείπα. Γιατί δημιουργήθηκε η διεύθυνση αυτή. Ως εργαλείο για την εφαρμογή της θέλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχειριστεί κρίσεις με μεγαλύτερη ακριβώς συνέπεια. Α, μου διόρθωσαν το όνομα, ευχαριστώ πολύ. Για να συνδυάσουμε το στρατιωτικό με το πολιτικό σκέλος. Η διεύθυνση λοιπόν αυτή συνδυάζει την παλαιότερη διεύθυνση που διαχειριζόμουν που ασχολούνταν μόνο με στρατιωτικά και την ανάλογη διεύθυνση για τα πολιτικά. και έτσι συνδυάζονται, συνεργάζονται πολλά στρατιωτικά αρχηγεία κρατών της Ένωσης τουλάχιστον στην πρώτη φάση του στρατηγικού σχεδιασμού. Τα δύο πλέον εκτήματα που διαθέτει μια τέτοια διεύθυνση είναι ότι αποτελεί ένα εργαλείο για την εφαρμογή και του σχεδιασμού μέσω αυτών των πολιτικοστρατιωτικών δομών και αυξημένες στρατιωτικές και πολιτικές δυνατότητες για τη διαχείριση των σχέσεων με τους εταίρους μας, των διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών με τις οποίες συνδιαχειριζόμαστε κρίσεις. Και επίσης τα στρατηγικά θόχματα και τα μαθήματα που παίρνουμε από τις επιχειρήσεις μας αναλύονται εκεί όλα τα οριζόντια θέματα όπως ανθρώπινα δικαιώματα και τα γέννη που παλαιότερα τα λέγαμε φύλλα. Αυτά όλα μαζί δηλαδή. Στρατιωτικά φύλλα. Και έτσι οι φραγμοί που υπήρχαν καταργούνται διότι παλαιότερα είχαμε εμπνευστεί από δομές άλλων οργανισμών της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπά, όπου υπήρχαν φραγμοί μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού σκέλους. Ενώ τώρα με τις νέες αυτές δομές συνδυάζονται τα δύο σκέλη. Και αυτό είναι κάτι το θετικό. Άλλο στόχος είναι να διασφαλίσουμε κάποια συνέχεια στην εφαρμογή των επιχειρήσεων, δηλαδή Εφόσον θεωρήσουμε ότι πρέπει να αρχίσει μια επιχείρηση είτε πολιτική είτε στρατιωτική, η ίδια δομή θα κάνει τον αρχικό σχεδιασμό και τις προβλέψεις μέχρι να καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης που να εγκρίνουν οι χώρες μέλη. Έτσι υπάρχει μεγαλύτερη συνέχεια στο σχεδιασμό των επιχειρήσεων και πολιτικών και στρατιωτικών. Επίσης, έτσι υπάρχει δυνατότητα στις επόμενες φάσεις να μπορεί να συνεχιστεί η παρακολούθηση αυτή των πραγμάτων με συνδυασμό και συνεργασία από άλλα όργανα όπως τα στρατηγία και αρχηγία των επιχειρήσεων και των σχεδιαστών της πρώτης φάσης. Η αρχική πρωτοβουλία θα το ξέρετε είχε ληφθεί από τη Γαλλική Προεδρία και τώρα μόλις άρχισε να εφαρμόζεται. Έτσι ώστε να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα η, εφαρμογή, η ταυτόχρονη εφαρμογή, η θέση ενισχύ της συνθήκης και των επιχειρήσεων αυτών. Με επικεφαλή στην κυρία Άστον. Σκοπός μας, επαναλαμβάνω για να καταλάβετε καλύτερα, είναι ο συνδυασμός και η ολοκληρωμένη διαχείριση των επιχειρήσεων που σχεδιάζουμε και που εγκρίνονται από τις χώρες μέλη. Είναι υπηρεσία που δεν θα αρχίσει βέβαια να λειτουργεί από αύριο, διότι ένας από τους στόχους της είναι ακριβώς να προβλέπει, να προσχεδιάζει θέματα για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων, αλλά ελπίζουμε να αρχίσει να λειτουργεί μέσα στο πρώτο εξάμεινο του επόμενου χρόνου. Αν έχετε απορίες βέβαια θα σας τις λύσω. Τώρα κάτι για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, το ζητήσατε και εσείς κύριε Πρόεδρε. Η επιχείρηση Αταλάντα σας είναι γνωστή γιατί συναντήσατε τον Ναύαρχο Χάντσον προηγουμένως νομίζω. την επόμενη εβδομάδα θα συμπληρωθεί ένας χρόνος από την αρχή της εφαρμογής της επιχείρησης αυτής καταπολέμησης της πειρατείας και θα λειτουργεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2010. Νομίζω ότι έχει αναγνωριστεί ότι η επιχείρηση αυτή είναι επιτυχής, διότι ανταποκρίθηκε στον ανθρωπιστικό της στόχο να συνοδεύει και να συνδυάζει προσπάθειες με το Διεθνές Επισητιστικό Πρόγραμμα για να βοηθάει τους πρόσφυγες στη Σομαλία. Έπειτα δημιουργήθηκε αυτό το κέντρο που που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν καλύτερες βέλτιστες πρακτικές και να ανταποκρίνονται στις επιθέσεις. Γιατί αυτές δεν αφορούν πάντοτε αποκλειστικά το κατά πόσον είναι επιχειρησιακά έτοιμη η στρατιωτική δομή, ε, φορούν και θέματα κλιματολογικών συνθήκων κλπ. Ένα σημαντικό στοιχείο της επιχείρησης αυτής είναι η στρατιωτική καθαρά ποιότητα της ναυτικής δύναμης που διαθέτουμε. Όταν η δύναμη αυτή συλλαμβάνει πειρατάς από την Κένια μέχρι τις Εχέλες πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να δίνεται μία δικαστική συνέχεια ώστε να φυλακίζονται τουλάχιστον οι πειρατέ εάν καταδικαστούν. Φροντίσαμε ιδιαίτερα οι συμφωνίες με την Κένια και τις Ειχέλες να σέβονται απόλυτα τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πέρα από αυτό, και ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε επιμείνει ιδιαίτερα, φροντίσαμε να αντιμετωπίσουμε και τις ρίζες της πειρατείας. Να δούμε δηλαδή τι θα μπορούσε να γίνει στην ίδια τη Σομαλία και ευρύτερα στην περιοχή της για να μειωθεί το φαινόμενο αυτό. Στη Σομαλία λοιπόν και στην περιοχή εκεί έχει αρχίσει να εφαρμόζεται μια ενωσιακή επιχείρηση ανάπτυξης και στήριξης διαφόρων παραγόντων διακυβέρνησης και απ' την άλλη επεξεργαζόμαστε μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Συμβουλίου για τη διαχείριση των κρίσεων φροντίζουμε να εκπαιδεύσουμε Σομαλούς στρατιώτες ώστε η μετάβαση σε μια τοπική καθαρά κυβέρνηση χωρίς βοήθεια να μπορέσει να γίνει όπως πρέπει. Να υπάρχει και μια στοιχειώδης ασφάλεια στο Μογκαντήσιο. Να υπάρξει μια εκπαίδευση λοιπόν των στρατιωτών της Σομαλίας μέχρι 2.000 Μελετήσαμε διάφορες πιθανές λύσεις. Όπως ξέρετε η Γαλλία στο Τζιμπουτί είχε ήδη κάνει μια πρώτη εκπαίδευση στρατιωτών. Τώρα θα κάνουμε μια εκπαίδευση και στην Ουγκάντα για διάφορους λόγους αλλά ιδιαίτερα γιατί η Ουγκάντα συνεισφέρει ιδιαίτερα στο άμισόμα και με τη βοήθειά του και της Αφρικανικής Ένωσης θέλουμε να εκπαιδευτούν στρατιώτες ώστε ώστε να είναι βέβαιο βέβαιο ότι θα πληρώνονται και ότι θα μπορέσουν να ενταχθούν σε μια σωστή στρατιωτική δομή για να ξέρουν ακριβώς πώς μπορούν καλύτερα να εξυπηρετήσουν τις αρχές που στηρίζουμε. Έτσι κατανέμουμε τις ευθύνες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχών της Ουγκάντας. Με στήριξη του Αμισόμ και της Αφρικανικής Ένωσης και φυσικά και του ΟΗΕ, καθώς και με ορισμένους άλλους εταίρους όπως τα Συνωμένα Πολιτεία που ήδη συνεργάζονται με την Ουγκάντα για την εκπαίδευση Σομαλών στρατιωτών. Τώρα για τις πολιτικές επιχειρήσεις πιο σύντομα θα σας τα πω και γιατί πιο σύντομα γιατί είμαι πρόσφατα διορισμένη και ο ρόλος της διεύθυνσής μου δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί ιδιαίτερα στο πολιτικό σκέλος. Το ΣΕΠΣΕΣΕ η θα τα καθορίσει αυτά σε δεύτερη φάση και επίσης είχατε και την περασμένη εβδομάδα πληροφορίες για τις πολιτικές αυτές επιχειρήσεις στην πρώτη συνάντηση της κυρίας Άστον σε δύο μέρες θα συζητήσουμε το Αφγανιστάν όπου είναι προφανές ότι πρέπει η επιχείρησή μας στο Αφγανιστάν να έχει όντως χαρακτήρα συμπληρωματικό με εκείνη του ΝΑΤΟ ώστε να προσφέρουμε κάτι παραπάνω. Επίσης θα έπρεπε να δούμε και ποιες, ποιες λέγω, τι πρέπει να κάνουμε για τη γεωργία. Ίσως καλό θα ήταν ε, να σχολιάσω και κάτι άλλο, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την μελλοντική μας δουλειά, δηλαδή οι ε, δυνατότητες που έχουμε, το δυναμικό διότι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Σουηδικής Προεδρίας ήταν να επεξεργαστεί ε, τις ε, συνέργειες μεταξύ του πολιτικού και του στρατιωτικού σκέλους. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχουν συνέργειες, αλλά πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες. Όπως σας είπα, ε, ένα εργαλείο αυτής της συνέργειας είναι και η συνεργασία και ε, για να μπορέσουν ε, να προσεγγίσουν οι ε, δυνατότητες οι πολιτικές με τις στρατιωτικές θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πολιτικές, ε, το πολιτικό δυναμικό δεν αναπτύσσεται με τον ίδιο τρόπο ή δεν αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με το στρατιωτικό σκέλος και θα πρέπει ε, για επιχειρήσεις στρατιωτικές ή πολιτικές όπως σε το χώρο, εις τη διοικητική μέρη, η στις αεροπορικές ε, μεταφορές, ε, ε, υπάρχει μια κοινή προσέγγιση. Αλλού όμως υπάρχουν διαφορές και χρειάζεται να γνωρίζει κανείς ποιες είναι αυτές για να συνεργαστούν οι δύο τομείς ε, παραδείγματος χάρη στον πολιτικό τομέα το κλειδί είναι να μπορούν να αναπτυχθούν ε, ε, στρατιωτικοί ή αστυνομικοί ή δικαστικοί με αποτελεσματικό τρόπο. Με τον Αλεξάνδερ Βάη, τον οποίο θα συναντήσετε μετά, εργαζόμαστε στα θέματα αυτά. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχόλησε και ε, ε, ε, επί του οποίου εστιάστηκε η προσοχή της τωρινής προεδρίας ήταν το θέμα των battle groups τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά έχουμε τα battle groups, αυτές τις μάχημες μονάδες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, διότι το πλαίσιο τους χρησιμοποιήσεως είναι περιορισμένο και συγκεκριμένο. Εάν δεν αναθεωρήσουμε λοιπόν αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει αρκετή ευελιξία για να μην χρησιμοποιούνται μόνο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο πενθήμερο τετράμινο, αλλά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν δύναμη ταχείας αντιδράσεως εάν το απαιτούν οι συνθήκες, κατά περίπτωση και με δύο βασικά στοιχεία, δηλαδή εάν συμφωνήσουν τα κράτη που καταρτίζουν αυτή τη μάχημη ομάδα, να μπορούμε να προχωρήσουμε αρκεί το Συμβούλιο να θεωρήσει ότι η χρήση των battle groups είναι ενδεδειγμένη για μια τέτοια κρίση. Ε, επίσης όσον αφορά τη συνεργασία με τους ε, διεθνείς ε, συνεργάτες μας το να έχουμε μία ευξημένη συνεργασία τόσο στρατιωτική όσο και πολιτική θα επιτρέψει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλύτερα με τις διεθνείς οργανώσεις. Παράδειγμα το ΝΑΤΟ, το οποίο στην προηγούμενη θέση μου γνώριζα καλύτερα από όλα. Ε, όταν έχουμε μεταξύ ε, επιτελείων ε, επαφές με τον ΝΑΤΟ ή όταν συμμετέχουμε στις υπουργικές συσκέψεις του ΝΑΤΟ. Όταν εγώ μιλούσα στο ΝΑΤΟ για επιχειρήσεις ήξερα ότι ε, ήμουν ε, σε άμεση σχέση αν πρόκειται για στρατιωτικά θέματα αλλά ε, σε έμεση αν μιλούσαμε για την πολιτική συμμετοχή όπου εμπλέκονται και τα κράτη-μέλη. Όταν λοιπόν θέλουμε να συνδυάσουμε το στρατιωτικό με το πολιτικό σκέλος για να αναπτυχθούν δυνάμεις η κατάσταση ήταν περίπλοκη γιατί υπάρχουν διάφορες, διαφορετικές απόψεις αλλά τώρα με το CNPD και την θέση του είπα του εκπροσώπου που είναι σε άμεση διασύνδεση μπορούν να υπάρξουν άμεσες συζητήσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Νομίζω το ίδιο μπορεί να ισχύσει για τις Ηνωμένε Πολιτείε, για την ε, Αφρικανική Ένωση ε, και για χώρους όπου εντάσσονται περισσότερο πολιτικές δυνάμεις και στον ΟΑΣΕ όπου υπάρχει συνεργασία με διάφορα κράτη. Αυτές λοιπόν είναι οι δραστηριότητες ε, τις οποίες αναπτύσσουμε ε, δεν θα επεκταθώ διότι αύριο θα συναντήσετε τη Lady Ashton και θα σας σχολιάσει ποιες είναι οι δυνατότητες που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας αλλά ήδη έχουμε φροντίσει ε, να αναπτύξουμε τις δομές που μπορούμε και οι διατάξεις ε, της νέας συνθήκης και οι διαθεσμικές διατάξεις θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε αυτή την συνέργεια και την αποτελεσματικότητα. Σας ευχαριστώ. Βλέπω ότι υπάρχουν διάφοροι συνάδελφοι που ζητούν το λόγο θα επανέλθω επειδή το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει πολύ στις επόμενες εβδομάδες και το οποίο έχουμε συζητήσει και προηγουμένως, δηλαδή το Αφγανιστάν και ε, πρέπει να αναρωτηθούμε ε, ποιος είναι ο στόχος της αποστολής ΕΠΟΛ που δυσκολεύεται να μπορέσει να ε, καλύψει τις υποχρεώσεις της, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της διότι το ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει μία training mission η οποία μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα γεωγραφικά και έχει ευρύτερους στόχους από την UPOL και ε, αναρωτιόμαστε εάν μπορεί κανείς να αναθέσει μία αποστολή σωστή στην UPOL η οποία να είναι λιγότερο αστυνομική και να αποβλέπει περισσότερο ε, την ανάπτυξη του δικαστικού πλαισίου ή στην εκπαίδευση και επιμόρφωση ε, των, ε, ε, των δικαστικών αντί των αστυνομικών διότι ε, ξέρουμε ότι στο Αφγανιστάν έχουμε πρόβλημα ε, πολιτικό σχετικά με το συντονισμό των δύο σκελών και ίσως θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα εντάξουμε την αποστολή ε, Ιούπολ στο πλαίσια του, των ευρυτέρων αποστολών και ε, συμφωνώ με τον Τιερή, ο οποίος ασχολείται με το Αφγανιστάν που τον ανησυχεί περισσότερο. Ο κύριος Γκαρτιέρη τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον Πρόεδρο για τη σχέση μεταξύ των αποστολών του ΝΑΤΟ, της Πολ και μια μεγαλύτερη συμμετοχή στην προσπάθεια οικοδόμησης θεσμών, ιδιαίτερα της δικαιοσύνης, ε, που είναι κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να γίνει στο Αφγανιστάν. Θέλω λοιπόν την άποψη της ευθύντριας της CMPD επ' αυτού. Που είπε και ο πρόεδρος Ντόνζο. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος το θεσμικό ζήτημα, τον ρόλο δηλαδή της νέας αυτής ε, υπηρεσίας CMPD. διότι αν δεν ε, παρενόησα, είναι πολύ σημαντική αυτή η θεσμική μεταρρύθμιση, επιφέρει μια πραγματική προστιθέμενη αξία. Πώς λοιπόν θα συνδυαστούν αυτές οι δραστηριότητες εφόσον στα πλαίσια των εξωτερικών πλέον δράσεων εμπλέκονται και όργανα που θεσμικά ανήκαν σε άλλες δομές. Ποια είναι η σχέση λοιπόν με την ε, στρατιωτική οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το στρατιωτικό επιτελείο, αλλά και την διακυβερνητική διαχείριση αυτών των θεμάτων στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ. Ε, oui, bonjour. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα το πρωί ε, και είναι μια ευτυχή ημέρα η 1η Δεκεμβρίου για την εφαρμογή της συνθήκης αυτής που χρειάστηκε τόσα χρόνια για να προχωρήσει δεν μπορώ καν να το πιστέψω ακόμη. Επανέρχομαι όμως σε αυτό που είπατε ότι οι πολιτικές αποστολές ε, έχουν πρόβλημα περισσότερο με το ανθρώπινο δυναμικό από ότι με τους στόχους όπως αναφέρατε το Αφγανιστάν, το Κωσιφόρ και σχεδόν όλες τις αποστολές. Άρα η ερώτησή μου είναι, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι καλή ιδέα να ξεκινά κανείς νέες αποστολές όπως στη Σομαλία ή θα έπρεπε καταρχήν να αναθεωρήσουμε και να ενισχύσουμε τις ε, ήδη ενεξελίξει αποστολές κατά τρόπον ώστε να μπορούν να στελεχωθούν με το προσωπικό το οποίο χρειάζονται. Φοβάμαι ότι διαφορετικά ε, υπάρχει ενδεχόμενο να διακινδυνεύσει η επιτυχία των εξελίξη ε, αποστολών, να ε, υπερβάλλουμε και να μην μπορέσουμε να καλύψουμε τον ευρύ χώρο τον οποίο προσπαθούμε να, στον οποίο προσπαθούμε να επέμβουμε και ουσιαστικά πιστεύω ότι θα πρέπει να να ε, μπορέσουμε να εστιάζουμε τη δράση μας για να ξεχωρίζουν και οι άλλοι συμμετέχοντες ε, μεταξύ ε, των στρατιωτικών και πολιτικών σκελών. Έχω και δύο ερωτήσεις. Καταρχήν η Ιράκ. Ποια είναι η επιτυχία αυτής της αποστολής αφού μετατέθηκε η αποστολή αυτή από τις Βρυξέλλες επιτόπου και υπό τη στις ισχύουσες συνθήκες εγκατελείφθηκε η ιδέα αυτή. Και δεύτερον στο Κονγκό, όπου νομίζω ότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται πραγματικά. Ε, κοιτάτε και αναθεωρείτε τους στόχους και τις εντολές των αποστολών μας, ιδίω στο Κονγκό δεδομένων των συνθήκων επιτόπου. Και γενικότερα θα ήθελα να ξέρω τι ε, πιστεύετε ε, για την κατάρτιση μίας λευκής βίβλου για την άμυνα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια πραγματική στρατηγική και προτεραιότητες ώστε τη μία φορά να μην ε, ο ένας προτείνει μία αποστολή από εδώ μια από εκεί και να υπάρχουν κριτήρια βάσει των οποίων θα αποφασίζει κανείς εάν θα ξεκινήσει μία αποστολή ή όχι, κυρία Μπράγκης. Θα ήθελα, θα ήθελα λέγω, θα ήθελα, όπως έλεγα λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι για τις δυνατότητες εκπαίδευσης θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Στην κεντρική Ευρώπη υπάρχουν χώρες που είναι μέλη και της Ένωσης και του ΝΑΤΟ, πρόσφατα μέλη του ΝΑΤΟ βέβαια και μερικές από αυτές δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες να συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της συμμαχίας λόγω του χαμηλού των ΑΕΠ. Πώς μπορούμε λοιπόν και εμείς να συμμετάσχουμε στις προσπάθειες της ως πλήρη μέλη διότι οι χώρες αυτές μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Άρα ως προς τη συμβολή του στον προϋπολογισμό πρέπει να δούμε και τι επαγγελματική δεοντολογία απαιτείται λοιπά, Μήπως το έχετε αναλύσει στο στρατό και την αστυνομία να υπάρξει κάποια μετεκπαίδευση των στελεχών στις χώρες αυτές για να φτάσουν και αυτές στο επίπεδο των υπολείπων ως προς το στρατό και την αστυνομία αν και διαθέτουν λιγότερα χρηματικά μέσα. Ευχαριστώ ο κύριος Πασκού. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως ε, θα μπορούσα να μιλήσω ρουμανικά, που είναι επίσης λατινογενής γλώσσα, αλλά θα περιοριστώ στα αγγλικά. Ε, εκτιμώ ιδιαιτέρως τη στιγμή κατά την οποία πρέπει να εναρμονίσετε, να ισοσκενιλήσετε τη συνέχεια και την διακοπή συγχρόνως διότι από τη μία πλευρά έχετε νέα άτομα, νέες δομές, νέες ευκαιρίες και τους προηγούμενους και όλα αυτά πρέπει να συντονιστούν και αντιλαμβάνουμε ότι είναι μία περίπλοκη στιγμή. Επίσης θα ήθελα να συμφωνήσω με όλους αυτούς οι οποίοι εξήραν το έργο του Σολάνα διότι άφησε το, ε, άφησε το σήμα του εις την πολιτική της Ευρώπης και ελπίζω ότι ε, θα μπορέσετε να ακολουθήσετε την ίδια πορεία και προς το μέλλον. Ε, προσωπικά διαβλέπω κάποια διαφορά μεταξύ της ε, διεθνούς εικόνας η οποία μετακινείται από τη διπολικότητα στην πολυπολικότητα όπου οι χώρες έχουν πολλές ευκαιρίες και τον πειρασμό να δράσουν ε, μονομερός και από την άλλη πλευρά έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας η οποία τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να κινούμεθα περισσότερο συλλογικά και από τη μία πλευρά λοιπόν ε, ε, αυξάνεται η συλλογικότητα και από την άλλη ε, πλευρά αυξάνεται και η πολυμερής αντιμετώπιση χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω υπό αυτές τις προποθέσεις πώς είναι δυνατόν να υποφεληθεί κανείς άμεσα από τις δυνατότητες που δίνει η συνθήκη της Λισαβόνης. Μήπως θα έπρεπε να περιμένουμε να ε, ε, αξιολογήσουμε καλύτερα ποιες είναι οι δυνατότητες που μας προσφέρει αυτή η συνθήκη προτού δράσουμε. Εσείς ε, πώς αξιολογείτε το θέμα. Επίσης διάβασα την στρατηγική της, ε, της, της Ισπανίας η οποία θέλει να μπλοκάρει τα σημεία κινήσεως των πειρατών και θα ήθελα να ξέρω πώς αξιολογείται αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. πρόληψη της κρίσεως θα πρέπει να αναφέρεται αυτή η υπηρεσία που διευθύνεται. Και το λέω αυτό διότι είναι προφανές ότι έχετε κατά νου κάποιες ε, περιοχές του κόσμου όπου, όπου υπάρχουν πολλές ανησυχίες Από την πλευρά της πρόληψης, ποιες είναι οι περιοχές του κόσμου που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής σας. Η κυρία Γενική Διευθύντρια, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για τα πολύ σημαντικά σας ερωτήματα. Δύσκολα όλα, και επί της ουσίας. Γι' αυτό είναι και σημαντικά εξάλλου. Για το Αφγανιστάν. Ναι, ναι λέγω. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αποστολή Γιπόλ σε σχέση με αυτά που αποφάσισε το να το πλέον να κάνει πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο περισυλλογής και νομίζω ότι θα είναι ένα από τα πρώτα θέματα που θα εξετάσει η κυρία Άστον. Γιατί αντιμετωπίζουμε αυτές τις δυσκολίες. Και αφορά αυτό που ρώτησε και η κυρία Ρόντερ. Υπάρχει δυσκολία αναδίπλωσης του προσωπικού στα πλαίσια μιας μη στρατιωτικής παρέμβασης. Η αστυνομία, η δικαιοσύνη δημιουργείται για να καλύψει εσωτερικές ανάγκες με ένα προϋπολογισμό και κάποιους πόρους που έχουν προβλεφθεί για την κάλυψη των εσωτερικών αναγκών Έναντι της ε, δημοσιονομικής καταστάσεως ε, και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλά είναι πολύ δύσκολο να στείλουμε στο εξωτερικό αστυνομικούς ή δικαστές. Είναι δύσκολο να στείλουμε οποιονδήποτε, όχι μόνο αστυνομικούς και ε, δικαστές, αλλά το θέμα της, των ανθρώπινων πόρων είναι πιο σημαντικό ως πρόβλημα από ότι ο εξοπλισμός, ελικόπτερα ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, αστυνομικοί και δικαστές πάντα χρειάζονται, ενώ στρατιώτες, όταν δεν υπάρχει πόλεμος, περισσεύουν ούτως υπήν και μπορούν να αποσταλούν πιο ευκόλως. Και για το Αφγανιστάν, όντως αντιμετωπίζουμε δύο πρόσθετα προβλήματα Πρώτα απ' δεν υποστηρίχτηκε η αστυνομική αποστολή μας από το ΝΑΤΟ στρατιωτικά. Δεν εξευρέθη συμφωνία λοιπόν για τον σχεδιασμό αυτής της υποστήριξης παρόλο που προσπαθεί ε, το επιτελείο του ΝΑΤΟ να το επιτύχει. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα παραπληρωματικότητος με τον ΝΑΤΟ. Μίλησα για παραπληρωματικότητα. Υπάρχει, πιστεύω. Στις επαφές που έχουμε με το ΝΑΤΟ και στο στρατιωτικό και στο μη στρατιωτικό επίπεδο ενδιαφέρεται το ΝΑΤΟ. Έχει αποδειχθεί ότι ενδιαφέρεται το ΝΑΤΟ για την εμπειρογνωμοσύνη που επιφέρει η αποστολή της ενώσεως στην Καμπούλ. Υπάρχει λοιπόν παραπληρωματικότητα, διότι μιλάμε για μια συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη που ε, μπορούμε να επιφέρουμε εμείς ως προστιθέμενη αξία για τους ε, Αφγανούς αξιωματούχους και λειτουργούς. Και στην Καμπούλ και σε άλλες αφγανικές πόλεις. πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν. Δεν μπορώ να προδικάσω το αποτέλεσμα στο οποίο θα καταλήξει η κυρία Άστον, αλλά μία από τις ε, εναλλακτικέ είναι να διευρύνουμε το φάσμα. και να επιτύχουμε μεγαλύτερη σύγκληση και συντονισμό με τον ΝΑΤΟ και στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στον ΝΑΤΟ δεν γνωρίζουν όχι μόνο τη συμμετοχή και την ενίσχυση που προσφέρουν τα κράτη-μέλη μεμονωμένα, αλλά ούτε καν η Ένωση στο σύνολό τη. Ο ρόλος της νέας υπηρεσίας και η θέση της στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Όπως γνωρίζετε, η κυρία Άστον είναι υπεύθυνη για τις δράσεις που θα προκριθούν δυνάμει της ΙΚΕΠΑ. Σε συνεργασία βεβαίως με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όμως έδωσε κάποιους προσανατολισμούς η οποία εις ό,τι αφορά τη διαχείριση των κρίσεων είτε για τη ΣΕΜΠΕΝΤΕ, είτε για το επιτελείο, το στρατιωτικό, είτε για τις ε, μη στρατιωτικές κρίσεις, είτε για το ΣΙΤΣΕΝ, γίνεται μια προσπάθεια εξορθολογισμού. το γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές καιροφυλακτούν και επαγρυπνούν πρέπει να αξιοποιηθεί. Και υπάγονται πλέον με άμεσο τρόπο στις αρμοδιότητες του του εκπροσώπου, της κυρίας Άστον. Νομίζω ότι με την νέα αυτή δομή τα πράγματα είναι πολύ πιο σαφή οι σχέσεις με την CPMD. με την ΚΕΠΑ ο σχεδιασμός είναι πιο σαφής. Εμείς κάνουμε τον στρατογικό σχεδιασμό, το επιτελείο το στρατιωτικό επιτελείο είναι αυτό το οποίο αποφασίζει για την εφαρμοσιμότητα ή μη της προτάσεως και μετά η ε, στρατιωτική, το στρατιωτικό σκέλος είναι αυτό που το εφαρμόζει αν χρειάζεται. Αυτή η δομή είναι πιο σαφής. Για την επιχειρησιακή ε, δράση είναι η ΣΕΠΕΣΕΣΕ αρμόδια και τελευταίο για το ΣΥΤΣΕΝ είναι η υπηρεσία που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αυτήν την ε, πλήρη εικόνα της πραγματικότητας που επικρατεί επί τόπου 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Είναι πολύ σημαντικός λοιπόν αυτός ο συντονισμός πριν λάβουν τις αποφάσεις του τα κράτη-μέλη. Γιατί τώρα άλλαξαν τα πράγματα. Όταν ε, λαμβάναμε μια απόφαση και λέγαμε θα κάνουμε μια πρέμβαση στο Κονγκό, στο Τσάντ, ε, μια στρατιωτική επιχείρηση, ξανά ήμουν εγώ υπεύθυνη, αλλά μόνο μέχρι ένα βαθμό, διότι μετά ήταν ξανά αρμοδιότητα της, ε, του στρατιωτικού σκέλους. Υπήρχαν λοιπόν πολλά κενά και τώρα ε, είναι πιο στεγανή ούτως υπήν η διαδικασία και υπάρχει μεγαλύτερη επικοινωνία για τις νέες αποστολές τώρα. Αυτό αν και αν αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ενδεχομένω σε άλλε αποστολέ. Θεωρητικά ναι, συγκεκριμένα όχι. Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση της Σομαλίας καθόλου. Στη Σομαλία θέλουμε να καταρτήσουμε τους στρατιώτες. Δεν είναι πολιτική η δράση. Δεν θα προσφύγουμε ούτε σε δικαστές, ούτε σε αστυνομικούς. Θα προσφύγουμε σε εκπαιδευτές σε στρατιωτικούς εκπαιδευτές. Αν προκριθεί αυτή η δράση, αν αποφασίσουν τα κρατημέλη να την ευλογήσουν, δεν έχει συμβεί αυτό ακόμα. Άρα είναι πολύ διαφορετικό από το Αφγανιστάν το θέμα αυτό. Θέλουμε στρατιωτικούς εκπαιδευτές να εκπαιδεύσουν στρατιώτες. Τώρα, στα πλαίσια της πιο γενικής προσέγγιση που έχουμε, δηλαδή να κάνουμε ίδιου είδους δράσεις και για τους αστυνομικούς και για τους δικαστές και για τους ε, δημόσιους ε, ε, υπαλλήλου. Αυτό είναι άλλο, άλλο ζήτημα. Διότι εμπλέκονται και άλλοι, η ΕΠΑ, η Αφρικανική Ένωση, είναι δική μας αρμοδιότητα να ασχοληθούμε με τα πάντα, με όλο το φάσμα των δράσεων και παρεμβάσεων. Μήπως υπάρχει κάποια οργάνωση ή κάποια δομή που να είναι σε καλύτερη θέση από εμά. Αλλά αυτό που θα πρέπει να διασφαλίσουμε είναι να μην υπάρχει σύγκρουση μεταξύ ε, της δικής μας δράσεως για την εκπαίδευση των στρατιωτών και άλλων ενδεχομένως δράσεων. Για το Ιράκ τώρα. Αν πρέπει να αναθεωρήσουμε την στρατηγική μας. Ζητώ μια πίστοση χρόνου. Ζητώ υπομονή, διότι... Ναι, είναι προφανές, είναι προφανές ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει, αλλά δεν είμαι έτοιμη ακόμα να απαντήσω. Δεν είμαι έτοιμη. Est-ce qu'il est qu y a euh, Τώρα, Μήπως χρειάζονται διαφορετικές δομές, μία για την στρατιωτική και μία για την μη στρατιωτική παρέμβαση. Χρειάζονται και τα δύο. Αλλά με επικοινωνία, με διαλειτουργικότητα. Το ίδιο και για τις επιχειρήσεις. Στα, στο στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού θα πρέπει να διαρωτηθούμε από όλο το φάσμα των μέσων που έχουμε στη θέση μας ποιο είναι το πλέον κατάλληλο. Πάτε για παράδειγμα τη γεωργία. Τον Αύγουστο πέρσι δεν ξέραμε ακριβώς τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ξέραμε ότι θέλαμε να κάνουμε κάτι αλλά το Συμβούλιο δεν γνώριζε στις 13 Αυγούστου τι θα έκανε. Θα ήταν μια παρέμβαση μη στρατιωτική. Θα ήταν μια παρέμβαση στρατιωτική. Το μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας έχει ευρύτερο φάσμα. Έχει και στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα. Τον Αύγουστο δεν ξέραμε. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία, επικοινωνία, αλλά μετά έρχεται ένα άλλο στάδιο όπου συμφωνώ μαζί σας ότι τα πράγματα ξεκαθαρίζουν και θα πρέπει να σεβαστούμε την α, ιεραρχία που υπάρχει σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του στρατιωτικού τομέα και του μη στρατιωτικού τομέα. για το Κονγκό. Υπάρχουν δύο αποστολές, η στρατιωτική και η μη στρατιωτική. Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών στις οποίες προσκρούμε και το έχουμε συζητήσει και στα Ηνωμένα Έθνη για τη συμπεριφορά του στρατού που υποστηρίζουμε. Βία, βιασμοί κτλ. Η ΟΝΟΚ έχει ενσκύψει επί του θέματος και θέλουμε να ολοκληρωθεί το σεξ στο Κονγκό αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα διότι εξαρτάται και από τη θέση του Πρόεδρου Καμπίλα και της επιτόπου πραγματικότητος. Λευκή βίβλος white book όπως λέμε στα γαλλικά. Προσωπικά εκφράζομαι πάλι διότι ε, την αίσθησή μου προσπαθώ να σας μεταδώσω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επίσημη θέση από αυτό. Υπάρχει η στρατηγική ασφαλείας. Η στρατηγική ασφαλείας, λέγω, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της έχουμε ασχοληθεί. Τώρα, αν θα πρέπει στο Συμβούλιο να ξεκινήσει μια διαδικασία, ένα εγχείρημα τύπου λευκής βίβλου, white book, για να συνεννοούμαστε, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Διότι η έννοια της λευκής βίβλου ε, έχει διαφορετικό περιεχόμενο από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Είναι πάντως ένα είδος στρατηγικού σχεδιασμού το ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει συγγνώμη, ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Υπάρχει αυτή η στρατηγική της ασφάλειας. Να ξεκινήσουμε τώρα εμείς το δικό μας. Ε, δεν ξέρω αν θα ήταν σωστό. Έχουμε και τα headline goal, όπως λέμε, που καθορίζουν πολύ το περιεχόμενο των δράσεων και τις προτεραιότητές μας. Οπότε η δική μου ε, αίσθηση είναι ότι εφόσον υπάρχει στρατηγική και εφόσον υπάρχουν και τα headline goal, θα πρέπει από αυτόν να επικεντρωθούμε εις ό,τι αφορά τις ε, φιλοδοξίες μας. Στρατιωτικός τε και πολιτικός πώς. Υπάρχουν πολλά επιτάπητος και θα πρέπει να τα συνδυάσουμε. Και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μέσο πρόθεσμους και όχι βράχη πρόθεσμους στόχους. Για την εκπαίδευση, για την κατάρτιση. Ε, είναι πολλά τα στοιχεία που καλύπτει ο όρος αυτός. Υπάρχει μια γενική κατάρτιση με την συμμετοχή του κολεγίου πολιτικών και στρατιωτικών δράσεων με τη συμμετοχή αστυνομικών, στρατιωτικών, διπλωματικών, αξιωματούχων Θέλουμε το δικό μας πρόγραμμα κατάρτισης να επικοινωνεί καλύτερα με το κολέγιο, την αστυνομική ακαδημία και όλα αυτά θα πρέπει να συγκλίνουν και θα πρέπει να κινηθούμε σταδιακά, διότι τίθενται και σοβαρά δημοσιονομικά ζητήματα πόρων και βεβαίως θέματα εκπαίδευσης πριν την μεταγωγή των εκπροσώπων μας ε, στα πλαίσια της αποστολής επιτόπου. Τώρα εντέθη ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά την βούληση και την διάθεση των κρατών μελών να συνεργαστούν και να δράσουν από κοινού. Είναι πολιτικό. Είναι άκρος, άκρος, άκρος πολιτικό το ζήτημα και νομίζω θα το αφήσω στην ε, κυρία Άστον, την ύπατη εκπρόσωπο να ε, το σχολιάσει. Εγώ πιστεύω ότι η νέα συνθήκη μας δίνει τη δυνατότητα να δράσουμε καλύτερα. Είναι ένα καλύτερο μέσο. Είναι ένα καλύτερο μέσο, επαναλαμβάνω. Έχουμε νέες ευθύνες και νέες δυνατότητες. Και έχουμε και τη δυνατότητα να υποβάλουμε προτάσεις πλέον. and to encourage them thus by being a proper structures, professional, on which they can rely. Um, On the the question... Για το ερώτημα των επιχειρησιακών μας επιτελείων θα το σκεφτώ και θα απαντήσω αργότερα. As regard the, your, your last question about uh, crisis prevention. ό,τι αφορά την πρόληψη των κρίσεων. Η νέα δομή, η CMPD, θα είναι κομμάτι της νέας διευρυμένης υπηρεσίας, της νέας διευρυμένης δομής στα πλαίσια της γραμματείας. Νομίζω ότι μπορούμε έτσι να συνεισφέρουμε στην πρόληψη των κρίσεων αποτελεσματικότερα. Αλλά αυτό το έργο είναι κυρίως και κατά πρώτο λόγο πολιτικό. Πολιτικό. Η Χέλγα Σμιτ, ο Ρόμπερτ Κούπερ, η πρόληψη των κρίσεων αφορά τη διαμεσολάβηση κτλ. Είναι και αυτό θέμα κυρίως πολιτικό. Και μετά είναι η προετοιμασία μιας στρατηγικής και αυτό κυρίως πολιτικό μέλημα. Σε ορισμένε περιπτώσει μπορούμε να βασιστούμε σε κοινοτικά μέσα και όργανα. στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Αλλά θα έλεγα γενικά για την πρόληψη ο ρόλος μας είναι κυρίως βοηθητικός. Ευχαριστώ πολύ κυρία Διευθυντή. Μήπως θέλει κανένα συνάδελφος να σχολιάσει ή να θέσει καμιά απορία του. Ε, τότε σας ευχαριστούμε. Όπως είπατε, τώρα πρέπει ο ύπατος εκπρόσωπος να τα λύσει ορισμένα από αυτά τα θέματα. Αύριο στην ΕΠΕΞ θα γίνει μια ακρόαση με την κυρία Άστον. Ιδιαίτερα για το πώς θα διασυνδεθούν όλες αυτές οι υπηρεσίες, ούτως ή άλλως νομίζω καλό θα ήταν να ξανάρθετε να μας δείτε μετά από μερικούς μήνες για να έχετε κάποια μεγαλύτερη εμπειρία στην διαχείριση της διεύθυνσής σας. Πάντως σας ευχαριστώ και για τη σημερινή σας προσέλευση, την ιδιαίτερη αυτή ημέρα της αποχώρησης του Χαβιέρ Σολάνα και της θέσεως ενισχύει της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα δούμε αν θα οργανώσουμε και καμιά γιορτούλα για την αποχώρησή του. Θα περιμένουμε τώρα λίγα λεπτά μέχρι να προσέλθει και ο κύριος Αλέξανδρος Βάης, Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξαναξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας για την κάποια καθυστέρηση και με μεγάλη χαρά θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Αλεξάνδρ Βάης, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο ε, Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑ και θα μας παρουσιάσετε τις λειτουργίες, τις αρμοδιότητες και τις επιχειρήσεις και αποστολές τις οποίες διευθύνεται γιατί είμαστε νέοι στο Κοινοβούλιο και δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις αρμοδιότητές σας και μετά θα περιμένουμε να μας εξηγήσετε τις τελευταίες εξηγήσεις, να μας δώσετε τις τελευταίες πληροφορίες ε, με τον ε, νέο ο Διευθυντή Αμήνης ε, και σχετικά με τη συζήτηση που είχατε προσφάτως και θα έπρεπε ίσως να διερευνήσουμε για τον οργανισμό σας τι σημαίνει να εργάζεστε στο νέο πλαίσιο της Συνθήκης Λισαβόνας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Κύριε Ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή την συνεδρίαση της Υποεπιτροπής σήμερα και είναι η, πρώτη μου παρουσίαση μετά από την εκλογή του νέου Ευρωκοινοβουλίου ε, και ε, θέλω να χαιρετήσω την συνεργασία μου που είναι η πρώτη με την Επιτροπή σας και ελπίζω ότι θα τα λέμε και στη συνέχεια. Σήμερα το, η συνθήκη της Λισαβόνας άρχισε να ισχύει και αυτό ε, επηρεάζει και τον οργανισμό μας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας υπό την ηγεσία της κυρίας Κάθριν Άσον και οι Υπουργοί Αμήνης έλαβαν πολύ σημαντικές αποφάσεις στις 17 Νοεμβρίου σχετικά με τις ε, προβλεπόμενες δράσεις για το 2010. Θα ασχοληθώ με τρία θέματα Καταρχήν ε, το, την γενική κατάσταση τη, του ΕΟΑ μετά από πέντε χρόνια λειτουργίες θα αναφερθώ ε, στα επιτεύγματα και στις δυνατότητες που διαβλέπουμε για το μέλλον και στη συνθήκη της Λισαβόνας και της επιπτώσεις της ε, στον οργανισμό. Καταρχήν πρέπει να σας πω ποια είναι η ισχύουσα κατάσταση. Είχαν υπάρξει πολλές αφιβολίες για την επιτυχία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και πίστευαν ότι ε, θα αποτελέσει ένα γραφειοκρατικό εργαλείο στα χέρια των εμπειρογνωμόνων, το οποίο θα αγνοούν εννοούσαν οι πολιτικοί. Δεν συνέβη όμως αυτό, διότι σιγά σιγά οι Υπουργοί Άμυνας ε, ενεπλάκησαν εις ε, την λειτουργία ε, του οργανισμού, τον στήριξαν και παρόλο που το ότι ένας τέτοιος οργανισμός με 100 υπαλλήλους δεν θα παραήγαγε τίποτα, έκαναν λάθος και η επιτυχία οφείλεται στο μικρό μέγεθος. Είμαστε ε, ρεαλιστές ε, και καθόλου γραφειοκρατικοί και ε, αναγνωρίζεται η προσήλωσή μας στην καλύτερη δυνατή απόδοση υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί, ο, το ΝΑΤΟ, ο, ε, πολλοί άλλοι και εμείς αποδείξαμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε συνδυάζοντας τις στρατιωτικές ανάγκες, την έρευνα, την τεχνολογία, την αγορά και ε, ε, την ε, ανάπτυξη ε, τεχνολογικών δυνατοτήτων. Επενδύουμε ιδίως στην έρευνα και γι' αυτό μετά από πέντε χρόνια είμαι αρκετά αισιόδοξο και υπερήφανος διότι οι μέτοχοί μας στα κράτη δηλαδή έχουν ενισχύσει την ε, συμμετοχή τους συνεργαζόμαστε με την ε, ΟΚΑ, την ε, Ευρωπαϊκή, ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος στη Βόνη και με τα κράτη-μέλη και επιπλέον αυξήθηκε το ενδιαφέρον των τρίτων χωρών για να συνεργαστούν μαζί μας και να συμβάλλουν στα προγράμματά μας. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Και τέλος έχουμε αρχίσει ε, με ένα ουσιαστικό διάλογο εκ του σύνεγγις με το Πεντάγωνο στην Αμερική και προσβλέπουμε στα αποτελέσματά του. Τίποτα όμως δεν είναι δεδομένο. Θα συνεχίσουμε να ε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις δυνατότητές μας, να έχουμε πιο στενή τεχνολογική και ερευνητική συνεργασία, να προωθήσουμε τα προγράμματά μας και ε, να ανοίξουμε την ε, ε, αγορά της άμυνας στην Ευρώπη και να ε, την τοποθετήσουμε σε καλύτερη βάση. Οι κλιματολογικές αλλαγές δεν είναι ο εχθρός μας, διότι τα κράτη πρέπει να συνεργαστούν διασυνοριακά και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Συνεργασία θα λύσει το πρόβλημα. Τώρα έρχομαι στο δεύτερο μέρος της παρεμβάσεως μου σχετικά με τα μεγάλα προγράμματα. Το να ε, λύσουμε την ανεπάρκεια των ελικοπτέρων είναι ένα από τα ε, προβλήματά μας και στις 17 Νοεμβρίου ε, αποφάσισαν οι Υπουργοί να ξεκινήσουν ένα νέο πρόγραμμα HDP με δύο ασκήσεις και ένα εκπαιδευτικό συμπόσιο το χρόνο και θα μπορέσει ο οργανισμός αυτός να αναπτύξει τις δυνατότητές μας, διότι πολλές φορές δεν χρειάζεται ε, μεγάλη οικονομική συνεισφορά για να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες. Πέραν αυτού ασχολούμαστε με ε, ε, τα οχήματα εις το κανονικό διάστημα χωρίς να είναι επανδρομένα και ε, προσπαθούμε να τα προωθήσουμε και τεχνολογικά και βιομηχανικά για να χρησιμοποιηθούν και ε, στον πολιτικό τομέα ή στο μέλλον για την ε, παρακολούθηση της ναυτιλίας και του εναερίου χώρου ε, μπορούν να παρακολουθήσουν επίσης τι άλλο πετάει γύρω τους και η ADA έχει ε, υπογράψει μία συμφωνία με το πρόγραμμα MITCAS για την ανάπτυξη της τεχνολογίας αισθητηρίων και κενών, δηλαδή ε, να μπορέσει να αποφύγει, μάλλον αισθητηρίων προς αποφυγή για να αποφύγουν τις ε, συγκρούσεις στον αέρα. Το πρόγραμμα αυτό θα προχωρήσει μέχρι το 2012 και έχει προσελκύσει στο ενδιαφέρον και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα άλλο βασικό θέμα είναι το πλαίσιο συνεργασίας για να αυξήσει τις συνέργειες από πλευράς πολιτικής ασφαλείας, διαστημικής συνεργασίας και ε, με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος θέλουμε να καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο οι τρεις εμπλεκόμενοι οργανισμοί θα συγχρηματοδοτήσουν και ε, θα συνεχίσουν να ελέγχουν τους πόρους τους. Παραδείγματος χάρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, θα ελέγχει τους, ε, τη χρηματοδότηση που προσφέρει αλλά θα μπορούν και οι τρεις θεσμοί να υποφεληθούν από την κοινή αυτή χρηματοδότηση και θα μπορέσουν να αναπτύξουν δίκτυα για να ε, βελτιώσουν την παροχή πληροφοριών ε, θα ε, εξεργαστούμε περισσότερο τις λεπτομέρειες και ε, θα ε, διατυπώσουμε προτάσεις μέχρι τέλος ε, Απριλίου 2010. Έχουμε το θέμα του στρατηγικού airlift, δηλαδή μεταφοράς και παραδόσεως δια του αέρα θα μπορούσα να σχολιάσω πολλά προγράμματα αλλά θα χρειαζόμουν πολύ καιρό και γι' αυτό τώρα έρχομαι στο τελευταίο μέρος δηλαδή πώς η συνθήκη της Λισαβόνας επηρεάζει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας όπως ξέρετε ε, να βαθμίζεται ο οργανισμός ιδίως στα πλαίσια της κοινή ε, πολιτικής άμυνας και στρατηγικής και ε, το πρώτο στόχος είναι να διαπιστώσουμε ε, ποιες είναι οι ανάγκες και να επιβεβαιωθούν οι ανάγκες αυτές μέσω αποφάσεως του Συμβουλίου, διότι ήδη πέρυσι είχαμε συμφωνήσει ότι ε, βάσει της αποφάσεως του Συμβουλίου του, της 12ης Εβδόμου 2004 θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και είναι πολύ βασικό ότι η κοινή δράση δεν θα αμφισβητηθεί διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργούσαμε ε, ε, μακροσκελής ε, διαπραγματεύσεις ενώ τώρα έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχει μία συνεχής δομημένη συνεργασία και οι χώρες οι οποίες έχουν υψηλότερα κριτήρια και έχουν δεσμευτεί αμοιβαία ε, για πιο φιλόδοξες αποστολές θα μπορέσουν να προχωρήσουν ε, ως μία μικρή ομάδα και ε, η συνθήκη θα αξιολογεί τις συνδρομές των κρατών μελών και ο οργανισμός θα αναφέρεται άπαξ του τους στο Συμβούλιο κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει και να εφαρμόσει τις συστάσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου. Άρα θα αποτελέσει ένα ε, στοιχείο ουσιαστικό της δομημένης συνεργασίας αλλά, θα, ε, επιτρέπει επίσης ε, την κατάρτιση του οργανισμού αυτού. Η επιλογή των μελών είναι πολιτική, αλλά τα βασικά θέματα για μας είναι ότι θα πρέπει ο οργανισμός αυτός να βασίζεται στις δυνατότητες του, να μπορέσει να είναι όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε η Ευρώπη να καταρρεύσει σε διάφορες ομάδες εκ των οποίων άλλοι θα ηγούνται και άλλοι θα σέρνονται ε, πίσω. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα ε, μεταβλητής γεωμετρίας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον σαν βάση για μια ευέλικτη και ουσιαστική συνεργασία διότι θα πρέπει να βασιθούμε ε, εις τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και να θα εξετάσουμε αν χρειάζεται μόνο μία μόνιμη ε, δομή ή πολλές. Τα ερωτήματα αυτά δεν μπορεί να τα απαντήσει μόνος του ο Οργανισμός Άμυνας ε, ο οποίος ουσιαστικά αποβλέπει σε μια παραγωγική συνεργασία και καταλήγω λέγοντας ότι μπορέσει κανείς, μπορεί κανείς να αποδώσει μόνο βάσει δομημένων προγραμμάτων και η θέλησή μας να συνεργαστούμε είναι το κλειδί της επιτυχίας. Η ε, ε, επιζήτηση συνεργειών είναι ένας ε, πολύ θετικός τομέας για τη συνεργασία των Βρυξελών με τα διάφορα θεσμικά όργανα και μεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών και τέτοιε συνεργασίε θα υπάρξουν σε επίπεδο όλων των κρατών μελών. Είμαστε ρεαλιστές, ε, ε, οικονόμοι και ε, προσπαθούμε να προωθήσουμε τα εργαλεία αυτά προς τα κάτι μέλη για να υποφεληθούν περισσότερο. Ε, είναι όλα αυτά επιχειρήματα για να υπάρχει πιο στενή συνεργασία αντί για το αντίθετο. Η συνεργασία καταλήγει εις ε, ε, την επιτυχία και γι' αυτό καλό την υποεπιτροπή να έρθει στον οργανισμό μας, να συναντηθεί μαζί μας και να συζητήσει οποιοδήποτε θέμα την ενδιαφέρει. Με τα μεγάλη χαρά θα σας δεχτούμε στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Βάης. Δεχόμαστε αυτή την πρόσκληση. Θα δημιουργήσουμε μια αντιπροσωπεία να σας επισκεφθούμε. Λοιπόν, πριν δώσω τον λόγο τώρα στους συναδέλφους, μια πορεια Συμμερίζομαι την εκτίμησή σας ότι η περίοδος αυτή κρίσης μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για την οργάνωσή σας γιατί με τις δημοσιονομικές δυσκολίες μπορεί να απαιτηθεί μεγαλύτερη συνεργασία. Απλά με τους αριθμούς που γνωρίζουμε δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται όλα αυτά προς τον δικό σας προπολογισμό που είναι 31 εκατομμύρια αν δεν απατώμε και δεν κατορθώσαμε μέχρι τώρα να τον κάνουμε πολυετή πράγμα που δυσκολεύει τον σχεδιασμό βέβαια και τον προγραμματισμό γιατί αυτός πρέπει να είναι μακροπρόθεσμος. Πώς εξηγείται αυτό και πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα εφόσον υπάρχει ακριβώς η κρίση η οποία απαιτεί περικοπές και στο δικό σας και σε άλλους προϋπολογισμούς ιδιαίτερα για την άμυνα. Λοιπόν, Περνάουζα Ευχαριστώ. Έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Μιλήσατε για τα προγράμματα ΚΕΤ 1 και ΚΕΤ 2. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι και ποιο είναι το κόστος τους. Η κυρία Κίστου Τροβόλ. Ευχαριστώ πολύ. για την παρουσίασή σας κύριε Βάιζ. Διάβασα το κείμενο. επανειλημμένο αναφερθήκατε στην έρευνα και στην τεχνολογία και θα ήθελα να μου πείτε πώς συνδυάζετε τις διάφορες δραστηριότητες έρευνας που απαιτούνται νομίζετε ότι μπορεί στο μέλλον να ενδιαφερθείτε περισσότερο για δραστηρι... ερευνητικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερα στα πλαίσια του 8ου προγράμματος, πλαισίου ακριβώς. Έπειτα, μιλήσατε για το κόμμα για τα ελικόπτερα. Σε ποια γλώσσα κάνετε την εκπαίδευση. Πρέπει όλοι να καταλαβαίνουν αγγλικά ή γίνεται εκπαίδευση και σε άλλες γλώσσες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ συγχαίρω για την παρουσίαση και ελπίζω ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας να λειτουργήσει με τρόπο ρεαλιστικό και όχι γραφειοκαρατικό ώστε να αποτελέσει παράδειγμα και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Could have huge implications. Ε, ε, έρευνα είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε να σώζονται ανθρώπινες ζωές. Αλλά από ό,τι ξέρουμε μάλλον οι Ηνωμένε Πολιτείε ασχολούνται με την εκτέλεση αποστολών στο Αφγανιστάν και αλλού. Η Ευρώπη έχει τέτοια ειδικά οχήματα ή οχήματα που να προλαμβάνουν τα ατυχήματα κατά την υπέρπτυση κατοικημένων περιοχών. Ευχαριστούμε. Πρώτος γύρος απαντήσεων. Ευχαριστώ. Το δικό σας ερώτημα ήταν το πιο προκλητικό, συγγνώμη για τους άλλους, αλλά οι διάφορες προοπτικές που υπάρχουν για τον προϋπολογισμό μας είναι πάντοτε το πιο ενδιαφέρον θέμα. Λοιπόν, για να δω το ιστορικό. Η ΕΟΑ, ο ΕΟΑ, από τις αρχές του το 2005 αποφάσισε να δημιουργήσει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο τριετές και προβλέπεται αυτό το τριετές πλαίσιο να το εγκρίνει με ομοφωνία το Συμβούλιο. Όχι με ενισχυμένη πλειοψηφία, αλλά με ομοφωνία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπορέσουμε να πείσουμε όλες τις χώρες μέλη. Μερικές όμως από αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική κρίση και πίεση, ιδιαίτερα για τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς και γι' αυτό έχουμε πρόβλημα. Έχουμε προσπαθήσει τέσσερις φορές να οργανώσουμε αυτό το τριετές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θα έλεγα ότι ο ΕΟΑ απέτυχε αλλά όλοι απέτυχαν και οι χώρες μέλη τέσσερις φορές να καθορίσουν ένα τέτοιο πλαίσιο. Όταν κατέφθασα πριν από δύο χρόνια στη θέση αυτή προσπάθησα να αναλύσω και να σκεφτώ γιατί απέτυχε τέσσερις φορές αυτό το τριετές δημοσιονομικό πλαίσιο και κατάλαβα ότι υπήρχαν πολλοί λόγοι. Πρώτον, δεν υπήρχε σωστή μέθοδος υπολογισμού των πόρων που θα χρειαζόμασταν για τα επόμενα τρία χρόνια. Κάναμε λοιπόν ένα τριετές πρόγραμμα εργασίας με πρόβλεψη για τους πόρους που θα χρειαζόταν, όχι μόνο χρήματα αλλά και ανθρώπινους πόρους. Για αυτούς δε Θέλησαμε να καθορίσουμε τι θα χρειαζόμασταν τα επόμενα τρία χρόνια και, σε αυτό το και πρώτη φορά φέτος καθορίστηκε αυτό το τριετές πρόγραμμα εργασίας. Επομένως φέτος είχαμε τη βάση για να κάνουμε τους υπολογισμούς μας, αλλά, αλλά υπήρχαν και άλλοι λόγοι για τη διαφωνία των χωρών μελών με τα προηγούμενα τριετή πλαίσια. Το τεχνικό πρόβλημα το λύσαμε δημιουργήσαμε μια σωστή βάση για τους υπολογισμούς, αλλά δεν λύσαμε ακόμα το θέμα της διαφοράς των πολιτικών απόψεων ως προς την ΚΕΠΑ και ΚΕΠΑ. Και φέτος κοντέψαμε να συμφωνήσουμε για αυτό το τριετές πλαίσιο, αλλά απλώς κοντέψαμε. Δεν υπήρξε ομοφωνία στο Συμβούλιο. Τι θα γίνει λοιπόν στο μέλλον. Θα ξαναπροσπαθήσουμε του χρόνου. Θα κάνουμε ένα καινούριο τριετές πρόγραμμα την άνοιξη του 10 και για την περίοδο 11 με 13 θα υποβάλουμε ένα πλαίσιο στις χώρες μέλη ως βάση για τον υπολογισμό θα υποβάλουμε ένα πρόγραμμα εργασίας για να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο χρηματοδοτικό. Θα συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας. Ο ΕΟΑ όμως δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της διαφοράς των πολιτικών απόψεων. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε για αυτό το θέμα είναι να είμαστε output oriented, ώστε να πείσουμε και όσους δεν έχουν ακόμη πιστεί. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν, output oriented. Το δεύτερο ερώτημα αφορούσε τις κατηγορίες α και β, τα, σχέδια, τα προγράμματα τύπου α και β. Αυτό έχει σχέση βέβαια με τη νομική βάση, δηλαδή το άρθρο 20 των κοινών δράσεων, όπου λέγεται ότι ο ΕΟΑ μπορεί να αναλάβει την πρωτοβουλία πρότασης συνεργατικών σχεδίων μεταξύ κρατών μελών, όπου μπορούν να συμμετάσχουν όλα. Αυτό είναι η κατηγορία Α. Οι χώρες που δεν ενδιαφέρονται για τέτοια προγράμματα μπορούν να εξαιρεθούν opt-out δηλαδή. Καλούνται όλοι να συμμετάσχουν και όσοι δεν ενδιαφέρονται μπορούν να εξαιρεθούν. Κατηγορία Α με δική μας πρωτοβουλία του ΕΟΑ. Κατηγορία Β είναι κάτι άλλο όμως. Δηλαδή η πρωτοβουλία, η πρωτοβουλία είναι των χωρών μελών. είτε μέσω διμερών ή πολυμερών πρωτοβουλειών για, ε, στα πλαίσια βεβαίως ε, της αρμοδιότητας της CDA και της ζητούν της CDA να εξεύρει άλλους συμμετέχοντες στην κοινή αυτή ε, επιχείρηση. Αυτές είναι οι δύο κατηγορίες ad hoc προγραμμάτων δυνάμει της δομής αυτής. Έρευνα και τεχνολογία πώς μπορούμε να συντονίσουμε καλύτερα τέτοιου είδους δραστηριότητε, είτε υφιστάμενες είτε αναφιόμενες και σε σχέση με το Ευρωμό πρόγραμμα πλαίσιο, ενδεχομένως και σε σχέση με το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο από το 2014 και εντεύθεν. Ανέφερα το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Συνεργασίας, European Framework cooperation. Περί τίνος πρόκειται, περί ενός συστηματικού τρόπου συντονισμού των προσπαθειών που αναλαμβάνουν η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, η ε, Επιτροπή ΓΔΕ Επιχειρήσεων και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αμήνης, βεβαίως με τη συμμετοχή των κρατών μελών. Να δώσω ένα παράδειγμα. τα UAB, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για λόγους φύλαξης των σύνορων. Ασφάλεια δηλαδή και όχι στρατιωτική δράση. Χρειάζεται όμως επιτελείο και έλεγχος. Κάποιος επιτόπου πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει, να διοχετεύει τις δραστηριότητες αυτής της ομάδος. Αυτό τον επιτελικό ρόλο τον χρειαζόμαστε και από πολιτικής και από στρατιωτικής απόψεως και μπορεί ακόμα και δορυφόροι να χρειαστεί να ελέγχουν την όλη διαδικασία. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να ενταχθεί στα πλαίσια του European Economic Cooperation. Η υπηρεσία διαστήματος μπορεί να διαχειριστεί θέματα που αφορούν τους δορυφόρους και τις δυνατότητες που έχουμε και εμείς με τα κράτη-μέλη για να βολιδοσκοπήσουμε τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν κάτι τέτοιο και να συνεργαστούμε και να συντονιστούμε βεβαίως και με, τους, και με τα δύο αναθεσμικά όργα. Να συμφωνήσουμε ας πούμε πνευματικά δικαιώματα στα συμβόλαια για την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων των ερευνών. Το χρήμα όμως δεν περνάει τα θεσμικά σύνορα. Δηλαδή, χρήμα από την Επιτροπή δεν πάει στην EDA. Χρήμα από την Υπηρεσία Διαστήματος δεν πάει στην Επιτροπή. Και ούτω καθεξής. συντονισμός και συγχρονισμός είναι αυτό που κάνουμε για να αποφύγουμε επικάλυψη προσπαθειών και για ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της έρευνας και τεχνολογίας. Για τις γλώσσες. Για το πρόγραμμα για κατάρτισης για τα ελικόπτερα. Είναι και μάθημα γλώσσας σε αυτό το πρόγραμμα. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα, ελληνικά, συγγνώμη, τα αγγλικά. Οπότε προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους συμμετέχοντες και από γλωσσικής απόψεως. Τώρα, για τις μελλοντικές τεχνολογίες, UAV, οι Υπουργοί ζήτησαν να εξετάσουμε την τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα UAV. Και αυτό διότι συνειδητοποίησαν ότι η πολιτική εννοώ, ότι η Ευρώπη δεν διδραματίζει κανένα ρόλο σε αυτήν την τεχνολογία. Οι πλατφόρμες αυτές είναι αμερικανικανικής κατασκευής και Ισραηλινής κατασκευής. Η Ευρώπη απουσιάζει <laughs> από το πεδίο αυτό το τεχνολογικό. Για τα UAV λοιπόν όταν θέλουμε να τα αγοράσουμε ο Ευρωπαίος φορολογούμενος πληρώνει και στρεφόμαστε κυρίως προς το Ισραήλ από αυτής της πλατφόρμας UAV αλλά από τα Υπουργεία Μήνης μας λάβαμε την εντολή να ξεκινήσουμε κάποιες σχετικές εργασίες για την ανάπτυξη κάποιας τεχνολογίας κλειδί που ουδής, ουδής στον κόσμο θα έχει μέχρι το 2012. Εμείς θα την έχουμε μόνο. Εμείς. Τα πέντε κρατημέλη που συνεισφέρουν στο πρόγραμμα αυτό θα έχουν αυτή την τεχνολογία. Και αυτό θα είναι κλειδί. Κλειδί για την μελλοντική θέση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο μέλλον. Ακόμα και οι Αμερικανοί εξέφρασαν ενδιαφέρον να ενημερωθούν. μα ζηλεύουν. Και αυτό νομίζω ότι θα συζητηθεί στα πλαίσια αυτού που ανέφερα προηγουμένως διάλογος EDA Πενταγώνου. Θα τους ενημερώσουμε, τους Αμερικανούς φίλους μας, και μπορεί να υπάρξει και κάποιο περιθώριο συνεργασίας, συντονισμού. Τα UAV e δεν θα πετούν μόνο στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, αλλά απανταχού του κόσμου, σε όλους τους εναέριους χώρους. Γι' αυτό τα πρότυπα νομίζω ότι είναι προς συμφέρον μας τεχνικές προδιαγραφές δηλαδή να αποτελέσουν αντικείμενο συντονισμού και συνεργασίας με τους Αμερικανούς. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό συνεργασία και οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται τα μάλα για τη δουλειά μας αυτή γιατί α, είναι ακριβώς αυτή η τεχνολογία που θα πρέπει να αναπτυχθεί. Ε, Τρει παρεμβάσει. Πρώτα ο κύριο Λαντσμπέργκη. Thank you, Chairman. Uh, may ask, uh, very... Ευχαριστώ. Απλά και ειλικρινά. Ερωτώ για τον εύξηνο πόντο και την βαλτική. Τι μπορούμε να κάνουμε για την αύξηση των δυνατοτήτων. Αν υπάρξει μία εξέλιξη από πλευράς ασφάλειας. Κάποιος τρελαθεί και κάτι κάνει. Είναι ένα ταχαίος μεταλλασσόμενο περιβάλλον. Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε. Ή μήπως θα περιμένουμε μόνο, θα περιμένουμε εννοώ μόνο να αναλάβουν πρωτοβουλία τα κράτη-μέλη πώς θα ανταποκριθούμε. Η ανταπόκρισή μας θα είναι κατηγορίας Α ή κατηγορίας Β. Ο κύριος Καλτέρη. molto interessante, molto completa. Ευχαριστώ πολύ πληρέστατη και άκρος ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας και συμφωνώ. Συμφωνώ με την άποψη ότι η EDA αποτελεί μεγάλη επιτυχία από τις πλέον σημαντικές των τελευταίων ετών. Μεγάλη λοιπόν επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία που δεν έχει εξαντληθεί, διότι έχει ακόμα μεγάλο περιθώριο εξέλιξης κάτι το οποίο καταδεικνύεται σαφώς νομίζω παρά τα προβλήματα που έχουμε τα οικονομικής φύσεως. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα ήθελα να επαναλάβω την υποστήριξη. Την υποστήριξη της ομάδος μας του Κοινοβουλίου. Γενικότερα πιστεύω στην υπηρεσία σας. Να αναπτυχθεί και να ανθίσει και να παγιώσει το έργο της. Και επί του προϋπολογισμού νομίζω ότι κάτι καλύτερο μπορούμε να καταφέρουμε. Τώρα, για τα PSC. Για την διαρθρωμένη συνεργασία. που αποτελεί ένα έμβριον μόνο, ένα πρώτον στάδιο με που θα οδηγήσει σε ένα έσχατο ενδεχομένο στάδιο, σε μια αγαστή επιχειρησιακή συνεργασία και αποτελεσματικότητα. Πώς θα το πράξουμε αυτό. Υπάρχει ένα δίλημα. Από τη μία δηλαδή η ελαστικότητα που απαιτείται, ελαστικότητα δηλαδή να χωρούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, στην προσπάθεια αυτή εννοώ και από την άλλη να υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας να υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας επιτόπου στις δράσεις αυτές. Αυτό θα σας ζητούσα να σχολιάσετε εις μεγαλύτερον βάθος. Δηλαδή μιλήσατε για μεταβλητή γεωμετρία. Όχι, εγώ θα μιλούσα για ομόκεντρους κύκλους. Αυτό είναι νομίζω σωστότερο εις ό,τι αφορά αυτές τις μορφές συνεργασίες. Και βεβαίως ζητώ και οποιοδήποτε άλλο επί σχόλιο αν έχετε, διότι η EDA θα πρέπει να υποστηρίξει αυτή τη μορφή συνεργασίας, αλλά και να εντοπίσει, να εντοπίσει λέγω, τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας αυτής. Αν έχετε να μας πείτε κάτι από αυτού, θα ήταν καλοδαχούμενο. Τέλος, κάτι για τις σχέσεις με το ΚΑΡ, που έχει διαφορετική φύση. Εξωτερική, να το πω έτσι. Το πλαίσιο αυτών των διαρθρωμένων επιχειρήσεων θα μπορούσε, και από αυτού ζητώ τη γνώμη σας, να συμπεριληφθεί εντός αυτής της νέας θεσμικής διάρθρωσης και οργάνωσης που έχουμε. Συμπληρωματικό της λοιπόν, αλλά και διαφορές μεταξύ CAR και EDA ή άλλων συναρμόδιων φορέων. Ευχαριστώ κύριε Μικολάη. Ευχαριστώ. Δύο μικρά ερωτήματα. Το επίγον του θέματος νομίζω την ευκαιρία που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Τώρα βέβαια υπάρχει και το θέμα της σπάνιδος πόρων. Μιλήσατε για κοινά ερευνητικά, συγγνώμη, επενδυτικά προγράμματα. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε περαιτέρω τη σκέψη αυτή για τις αναφιόμενες τεχνολογίες. Έχετε ήδη συμμετάσχει σε κάποιες προσπάθειες. Και το ΦΑΡ έχει κάποιους πόρους. Και το άλλο θέμα αφορά τις πληροφορίες, δηλαδή intelligence, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Τι γίνεται με τις πληροφορίες, intelligence. Υπάρχουν πολλοί τομείς Στου οποίου κατέχουμε υπηρεσίες και νομίζω ότι οι υπηρεσίες μας θα πρέπει να εκπαιδευτούν καλύτερα για να τις αξιοποιήσουν πληρέστερα. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ για την ε, ακριβή απάντησή σας. Ε, στην πρώτη ερώτηση όμως υπήρξε κάποια παρανόηση και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη και να διατυπώσω μία δεύτερη ερώτηση. Ε, αυτή τη στιγμή τι πρώτης και δεύτερης σειρά κατηγορίας προγράμματα υπάρχουν και ε, ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους έχετε διατυπώσει για την τρέχουσα περίοδο. Ευχαριστώ. Θα προσθέσω και εγώ μία ερώτηση για τις τρίτες χώρες, διότι αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα. Ήθελα να ζητήσω περισσότερες εξηγήσεις και επίσης εάν οι συνεργασίες τις οποίες έχετε με τις τρίτες χώρες προέρχονται μέσω του οργανισμού ή κατευθείαν μέσω ε, συνεργασιών που έχετε με εθνικούς οργανισμούς ή οργανισμούς κρατών μελών και βιομηχανίες κρατών μελών. Δηλαδή αν είναι συνεργασίες οι οποίες ε, μπορεί κατά περίπτωση να ε, αναπτύσσονται μεταξύ του οργανισμού και του εμπλεκομένου οργανισμού. Σας ευχαριστώ για τις ε, πολύ απαιτητικές σας ερωτήσεις. Ξεκινώ με την πρώτη. Πώς η EDA μπορεί να βελτιώσει ή αν βελτιώνει την δυνατότητα την ε, ε, αμυντική εις ε, την περιοχή της Βαλτικής και ποιες είναι οι δραστηριότητες για τη Μαύρη Θάλασσα. Στη Βαλτική έχουμε τρία κράτη που συμμετέχουν και βοηθούν πολύ την οργάνωσή μας. Και θα ήθελα να επιθυμίσω ότι μία από τις ε, δράσεις προτεραιότητας προέρχεται από το πρόγραμμα ανάπτυξης των ε, δυνατοτήτων, το οποίο θα εξηγήσω. Ξεκινάμε το 2006, όπου ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη ε, να μπορέσει ο ε, ΕΟΑ να ε, καθορίσει τις μελλοντικές απειλές για τις ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις αλλά και τα μέσα που θα χρειαστούν για να αντιταχθούν σε αυτές τις απειλές. Οπότε τότε αρχίσαμε να καταρτίζουμε στρατηγικό προγραμματισμό ε, και ε, το πρόγραμμα που ονομάσαμε ε, πρόγραμμα ανάπτυξης των δυνατοτήτων και του δυναμικού. Αυτό αυτό το πρόγραμμα παραδόθηκε στις 8 Ιουλίου 2008 ή στα κρατη και καταρτίζεται από, καταρχήν από μία παρουσίαση των βραχυπροθέσμων στρατιωτικών αναγκών ε, είναι η πτυχή Α και βασίζεται σε μία προβολή μέχρι το 2010 και σε έναν κατάλογο προόδου και καθορίζει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες. Το δεύτερο ήταν το Work Strand B δηλαδή ε, ο δεύτερος κύκλος εργασιών που ασχολείται με τις ε, απειλές και τις ανάγκες μέχρι το 2025, δηλαδή μακροπρόθεσμη αξιολόγηση, η οποία υιοθετήθηκε από τους ε, από τους Υπουργούς Αμήνης το 2006 στο Λέβι ε, και καλύπτει τις απειλές μέχρι το 2025 όπου αναλύσαμε τι χρειάζονται οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις για να αντιταχθούν σε αυτές τις απειλές. Και το τρίτο είναι μία βάση δεδομένων συνεργατική όπου ε, κάθε χώρα καταχωρεί τα ε, προγράμματα τα οποία οποία ξεκινούν και όπου θα μπορούσε να συνεργαστεί με άλλα κράτη-μέλη ε, και υπάρχει ε, και μία πτυχή για τα συμπεράσματα και τα μαθήματα που πήραμε από κάποιο πρόγραμμα και εδώ αναφερόμαστε εις ε, την ευθύνη του στρατιωτικού σκέλος το οποίο ε, καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με ε, το τι ουσιαστικά έγινε σε κάθε αποστολή και είναι ο έλεγχος της πραγματικότητος επί πραγματικών στοιχείων και έτσι καταρτίζεται το πρόγραμμα αυτό. Η πρώτη μορφή του προγράμματος ανάπτυξης ε, του δυναμικού ήταν ε, δοκιμαστική. Είχαμε όμως τονίσει ότι θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις. Μια από αυτές λοιπόν αυτές είναι ε, οι επιχειρήσεις με με ε, δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ε, ε, μία πρώτη προσπάθεια έγινε την άνοιξη του 2007 στο, στην Εστονία όταν κατέρευσε το σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δεν ξέρουμε ε, ποιος προκάλεσε αυτή την κατάρρευση. Είχαμε ορισμένες ιδέες, αλλά και πάλι η δυνατότητα να ε, προστατεύσουμε όχι μόνο στρατιωτικά, γενικότερα ε, τα δίκτυα υπολογιστών από προσβολές είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Και αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε υπό την ηγεσία του στρατιωτικού προσωπικού. Δεν ξέρουμε αν θα πετύχουμε ή όχι. Είμαστε ακόμη στα πρώτα βήματα και έτσι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Οι σχέσεις μας με την ΟΚΑ. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι με ρωτήσατε. Θεωρούμε ότι ο οργανισμός μας δεν είναι ένας οργανισμός διαχειριστικός αλλά ότι πρέπει να προκαλούμε τις και να διατυπώνουμε τις ανάγκες, να τις συντονίζουμε ε, να υπάρξει μία ερευνητική ε, δουλειά και ε, να αναπτύσσουμε τις, τα προγράμματά μας και να αναφερόμαστε στην έρευνα, στην παραγωγή και στην διοικητική μέρημνα όπως επίσης και στις δημόσιες αγορές. Δηλαδή δεν διαχειριζόμαστε επί καθημερινής βράσεως τα προγράμματα αυτά, αλλά υπάρχει με ένας άλλος οργανισμός διεθνής, ο οποίος είναι ήδη ε, κατευθυσμένος και μπορεί ε, να ε, διαχειριστεί τα προγράμματα αυτά ή όκα. Λοιπόν, το 2008 οι Υπουργοί Αμήνης Ευρωπαϊκής Ένωσης διακήρυξαν μέσω μιας διακήρυξης του Συμβουλίου ότι ο Οργανισμός Άμυνας και η ΟΚΑ ε, είναι προνομιούχοι συνεργάτες ε, εκ των οποίων ο ένας αναλαμβάνει τα προγράμματα στην φάση της κατάστασης κατάρτισης και ο ΟΚΑ στη φάση της ανάπτυξης και των δημοσίων αγορών. Ε, η ΟΚΑ λοιπόν είναι ε, ένας τρίτος οργανισμός με τον οποίο μπορούμε να έχουμε απλώς σχέσεις μέσω μιας διοικητικής συμφωνίας την οποία διαπραγματευτήκαμε φέτος, την παραδώσαμε στο Συμβούλιο και τώρα συζητάται στις επιτροπές του Συμβουλίου και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να τύχει τη στήριξη στο όλων των κρατών μελών πριν το τέλος του έτους εφέτος. Ε, τα προγράμματα κοινών ε, ε, επενδύσεων. Έχουμε δύο τέτοια προγράμματα. Το ένα έχει σχέση με την προστασία των δυνάμεων που ξεκίνησε το 2006 το, ε, μετά από απόφαση του 2003 ε, ξεκινήσαμε ε, να το χρηματοδοτούμε το 2007 και έχουμε ξεκινήσει το 2008 ένα δεύτερο πρόγραμμα κοινών επενδύσεων 15 εκατομμυρίων ευρώ που συμμετέχουν 15 κράτη-μέλη και το οποίο αναφέρεται στις μελλοντικές τεχνολογίες, δηλαδή σε ουσιώδη έρευνα και τεχνολογία. Έχουμε εντοπίσει Έχουμε εντοπίσει διάφορα θέματα διότι εκπαιδεύουμε αναλυτές οι οποίοι παρακολουθούν τις πληροφορίες οι οποίες διατίθενται και αναλύουν τους, τις δυνητικές απειλές. Όσον αφορά τα προγράμματα κατηγορίας Α και Β στο πρόγραμμα Intel, ε, δεν έχουμε δεν έχουμε ε, κανένα πρόγραμμα ούτε πρώτη ούτε δεύτερη κατηγορία σε αυτό το τομέα. Αλλά κάτι καταρτίζουμε και θα ήθελα να με βοηθήσετε σε αυτή την αναδυόμενη κατηγορία αλφα ε, ε, και στο πρόγραμμα το οποίο είναι δύσκολο να σας εξηγήσω Γι' αυτό θα σας παρουσιάσω μία λεπτομερή παρουσίαση των interface όταν θα έρθετε στις εγκαταστάσεις μας και θα σας παρουσιάσω και το πρόγραμμα αυτό. Η ερώτηση του Προέδρου σχετικά με τις ε, σχέσεις με τρίτες χώρες. Έχουμε καταρτήσει μόνο με μία τρίτη χώρα μία τυπική σχέση με την Νορβηγία που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά είναι ε, μέρος της WEAG η οποία διαλύθηκε και τότε ε, στη διάλυσή της είχαμε υποσχεθεί στην Νορβηγία ότι θα μπορεί να χαίρει διοικητικών συμφωνιών για να υποφεληθεί από τα προγράμματά μας. Και όντως το 2006 ε, ε, διατυπώθηκε αυτή η συμφωνία την οποία, ε, στην οποία συμφώνησε το Συμβούλιο. Το ίδιο έγινε το 2006 με την Τουρκία αλλά εκεί δεν στηρίχτηκε, δεν έτυχε της ομοφωνίας της στήριξης των του, μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και γι' αυτό δεν προχωρήσαμε. Τα κράτη-μέλη και οι τρίτες χώρες πρέπει να προσεγγίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους πολιτικούς ηθήνοντες, ε, τον είπα το εκπρόσωπο, το Συμβούλιο, να εκφράσουν την ε, ε, το ενδιαφέρον τους για να έχουν σχέση με τον ναι. Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Εμείς ε, σαν οργανισμός μπορούμε να έχουμε μόνο άτυπες σχέσεις, πράγμα το οποίο κάνουμε με τους Αμερικανούς, συζητάμε και με το Ισραήλ, ε, που ενδιαφέρονται επίσης για τον οργανισμό μας, αλλά πρόκειται απλώς για άτυπες σχέσεις. Αν κάποια στιγμή μπορέσουμε σε, στα πλαίσια αυτών των ατύπων συζητήσεων να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες ε, συμφωνιών με αυτά τα κράτη. Θα πρέπει να ε, υποβάλουμε την πολιτική αίτηση στους πολιτικούς ηθήναντες και να τους ζητήσουμε να μας επιτρέψουν να προσχωρήσουμε σε μία διοικητική συμφωνία. Αλλά ούτε η δυνατότητα στα τρία, στις τρίτες χώρες, ούτε αλλού δεν μπορεί να επηρεάσει αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λανσμπέργκης. Εγώ ακόμη περιμένω. Να μου πείτε τι γίνεται με τα Μιστράλ. Αντιλαμβάνομαι ότι αν όπως ε, στην ε, επίθεση κατά της Εστονίας το 2007, εάν κάτι συμβεί, θα πρέπει κάτι να υπάρξει, να υπάρχουν δηλαδή προληπτικά μέτρα για το μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι γίνεται σχετικά με την Βαλτική. Μας είπατε ότι υπάρχει μια ισορροπία σχετικά με την ασφάλεια στο βορρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως απλώς περιμένει τι θα συμβεί ή θα χρησιμοποιήσει τον ε, ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας για αντισταθμιστικά μέτρα. Παραδείγματο χάρη τα, βαλτικά, τα κράτη της Βαλτικής θα μπορούσαν να αποκτήσουν είτε τορπίλες είτε υποβρύχια ε, ή άλλες δυνατότητες κατά τρόπον ώστε όλες οι χώρες να μπορέσουν να επωφεληθούν από, τον, από την προσπάθεια ταχεία, τα, ε, ταχεία αφοπλισμού διότι τότε θα μπορούσαν να αναπτυχθούν καλύτερα και οι επιχειρήσεις οι σχετικές. Λοιπόν, εσείς πώς το βλέπετε, ποιο είναι το όραμά σας σαν Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας ε, απλώς αναλύεται εκ προημίου το τι πρόκειται να γίνει ή προχωράτε και παρακάτω. Ευχαριστώ. I try to explain. Θα προσπαθήσω να σας τα εξηγήσω. Αναλύσαμε μαζί με την Στρατιωτική Επιτροπή και το Στρατιωτικό Προσωπικό όλων των χωρών μελών, μαζί με αυτές και η Λιθουανία, τις απειλές μέχρι το 2025. Αυτό δεν το ανέλαβε μόνο ο ΕΟΑ, ήταν κοινή προσπάθεια του ΕΟΑ, της Στρατιωτικής Επιτροπής, του Στρατιωτικού Προσωπικού και όλων των χωρών μελών μεταξύ των οποίων και η Λιθουανία, Λετωνία και Εσθονία. Έχουμε λοιπόν μια σαφή εικόνα για τις πιθανές απειλές μέχρι το 2025 ή και 2030 ακόμα επιθέσεις ηλεκτρονικές ή όχι. Και αρχίσαμε ήδη να παίρνουμε μέτρα, αλλά αν η Λιθουανία ή άλλη χώρα μέλος της Ένωσης θέλει πληροφόρηση για να μπορέσει να λάβει μια εθνική απόφαση ως προς το πώς να αντιμετωπίσει μια απειλή, να έρθει να μας το θέσει, να συνεννοηθούμε. Και στις βαλτικές χώρες ισχύει αυτό και σε άλλες χώρες. Μπορεί να μην ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν, αλλά υπάρχει κάποιος. Εμείς δεν προτείνουμε σε καμία χώρα μέλος να αγοράσει ελικόπτερα από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία ή τη Γερμανία. Δεν εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Εμείς βοηθούμε τις χώρες μέλη να αναπτύξουν τις δυνατότητες που χρειάζονται. Εκείνες όμως θα παίξουν τον ενεργό ρόλο. Merci, Weiss. Ευχαριστούμε κύριε Βάις. Αν δεν υπάρχουν άλλες απορίες, σας ευχαριστώ για την εξηγήσει σας. Θα ξαναειδωθούμε για την δομημένη συνεργασία μόλις τα πράγματα γίνουν σαφέστερα. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας και σημειώνουμε την πρόσκληση να επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις σας. Τώρα θα ήθελα ο κύριος Κύρος Βόλσκι να έρθει εδώ για να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση των εργασιών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στην οποία είχε πάει μέσα Νοεμβρίου στο Εδιμβούργο. Donc, chers κύριος Κύρος Βόλσκι για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν αρχίσω, θα ήθελα να πω μία λόγια για το Εδιμβούργο. Να εξηγήσουμε γιατί είναι τόσο δυσαρεστημένος και ο πρόεδρος Λαντς Πέργκης. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι αν πρέπει να έχουμε κοινοτική άμυνα από τη μία και από την άλλη με μονομένες πωλήσει των προϊόντων. Εμείς θέλουμε τη συνεργασία για να αυξηθεί η ασφάλειά μας, αλλά αυτό συμβαδίζει με ατομικές αποφάσεις μεμονωμένες για τις πωλήσει όπλων από ορισμένε χώρες μέλη. Αυτό μπορεί να θέτει εν κινδύνο την ασφάλεια ορισμένων άλλων χωρών. Μπορεί ο κύριος Λάντς Πέργκης να μην είχε πλήρως καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει ή να τα είπε τόσο με τη συνηθισμένη του λεπτή ανάλυση και εμείς να μην καταλάβαμε. Λοιπόν, καταρχήν, η αντιπροσωπεία μας, της οποίας προείδρευα, πήγε στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ στο Εδιμβούργο πήγε 13 με 17 Νοεμβρίου. Αποτελούνταν από πέντε μέλη. Τάνοκ ήταν εδώ πριν. Πάσκου έφυγε. Κυρία Γκόμες και η κυρία Κράιζελ Ντέρφερ. Γενικά, δεδομένου του αριθμού αυτού που ήταν περιορισμένος, νομίζω ότι υπήρξαμε πολύ δραστήριοι. Το κυριότερο θέμα συζήτησης ήταν το Αφγανιστάν. Υπάρχουν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ εκεί, δεν είναι γνωστό. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε οργανώσει την συνάντηση. Φέτος 99 στρατιώτες της δύναμης αυτής σκοτώθηκαν και η δική μου χώρα είχε θύματα και γι' αυτό αφιερώθηκε η συνάντηση στη μνήμη όλων των ανατοϊκών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Η συνέλευση αυτή μοιάζει με το κοινοβούλιο στις αρχές του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του, δηλαδή αποτελείται από βουλευτές και από τις 28 χώρες. Και πολλές φορές είναι και οι ίδιοι, είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή. Στην Ολομέλεια και σε πέντε επιτροπές και συζητήσεις που οργανώθηκαν, εγώ ήμουν στην πολιτική αλλά προσπαθήσαμε η προσωπία να πάει σε όλες, συζητήθηκαν διάφορα θέματα της αρμοδιότητός των. Δηλαδή, κατά πόσον υπάρχει υποστήριξη της νατοικής αποστολής ή όχι από όλες τις χώρες και αν χρειάζεται περισσότερο περιφερειακή προσέγγιση όπως είπε η Ολομέλεια. Συζητήθηκε και ο ρόλος του Πακιστάν στην καταπολέμηση των διαφόρων εξεγέρσεων των Ταλιμπάν. Ο Ράσμουσεν προείδρευε στην επιτροπή στην οποία πήγα δεν θα σας πω λεπτομερώς ό,τι είπε, αλλά να σας αναφέρω μία φράση. Ζήτησε από τους κοινοβουλευτικούς να διαθέσουν περισσότερους στρατιωτικούς πόρους και άνδρες για την εκπαίδευση των Αφγανών στρατιωτών και είπε ότι αν τα παρατήσουμε και στρέψουμε τις πλάτες μας στο Αφγανιστάν τότε η Αλκάιντα θα επιστρέψει αμέσως. Ήταν εκεί και ο Ντέιβιτ Μίλιμπαντ που μίλησε στην Ολομέλεια και είπε ότι το Αφγανιστάν δεν πρόκειται να αποτελέσει έναν ατέρμονα πόλεμο, αλλά ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να λείπει από τις επιχειρήσεις. Επίσης, εκλήθησαν σκότι βουλευτές γιατί όπως ξέρετε το Εδιμβούργο βρίσκεται στη Σκοτία. Και ζήτησαν και αυτοί περισσότερους άνδρες να ασθαλούν στο Αφγανιστάν. Ο, υπήρχε και ο Καναδός βουλευτής Ζωάν ο οποίος ζήτησε απόσυρση το 2011 των Καναδών στρατιωτών και Γεωργιανοί που ζητούσαν περισσότερους άνδρες. Αλλά το κυριότερο συμπέρασμα ήταν ότι Αφού πήγαμε μαζί πρέπει μαζί και να φύγουμε. Άλλα θέματα. Η αναθεώρηση της στρατηγικής αντίληψης του ΝΑΤΟ ή η νέα στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ, κάτι σαν την ευρωπαϊκή στρατηγική αντίληψη, τις περικοπές των αμυντικών δαπανών, το Ιράν, από όπου είχε έρθει ο Άιον η Σομαλία, η τρομοκρατία, η πυραυλική άμυνα, η μη διάδοση και οι σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής με μια πολύ καλή παρουσίαση του στρατηγού Κλάους Νόρμαν. τους οποίους καλό στην ΕΠΕΞ και εδώ. Ήταν πολύ εμπνευσμένη η ομιλία. Α, η ομιλία του ήταν και πολύ ευρωπαϊκού χαρακτήρα, ευρωπαϊκού. Τι άλλα θέματα, η ασφάλεια των τροφίμων, η δημοσιονομική κρίση, οι κλιματολογικές αλλαγές. Μερικά μέλη εξέφρασαν αμφιβολίες ως προς το ρόλο του ΝΑΤΟ. Είχε συζητηθεί το κατά πόσο πρέπει να περιοριστούμε στο άρθρο 5 ή στις νέες στρατηγικές αντιλήψεις του ΝΑΤΟ. Οι ρωσικές λευκορωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στα σύνορά τους επίσης συζητήθηκαν και επ' αυτού το ΝΑΤΟ πήρε σαφέστατη θέση όπως μπορεί να ξέρετε, διαφορετική από τη δική μας. Τέλος, Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε ενδυνάμωση του διαλόγου με τον ΝΑΤΟ. Πρέπει να συμβάλλουμε πιο ενεργά στο διάλογο αυτό μέσω της συμμετοχής μας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ. Επίσης πρότεινα στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και ο ίδιος να πάει να επισκεφθεί το για να ενδυναμωθεί ο διάλογος. Πρέπει να έχουμε περισσότερες επαφές πάντως. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, την πρόταση αυτή σας την απευθύνω και σας να υπάρξει διάλογος με προσώπους του ΝΑΤΟ για να συμβάλλουμε και εμείς στην συγγραφή του νέου γράφου τουλάχιστον να ακούσουμε τα επιχειρήματα και να ακουστούν και τα δικά μας. Η Μαγδαληνή Ολμπράιτ μπορεί να έρθει γιατί έχει προσκληθεί ως μέλος της Ενδεκαμελούς Επιτροπής Σοφών του ΝΑΤΟ. Επίσης νομίζω ότι θα μπορούσαμε να εκμεταλλευθούμε το σημείωμα που έγραψε η Υπηρεσία Ενημέρωσης και Τεκμηρίωσης του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις μας με τον ΝΑΤΟ και την νέα του στρατηγική αντίληψη. Uh, into... Ιδιαίτερα στα θέματα που ενδιαφέρουν πολύ το ΝΑΤΟ Έχω προτείνει και δύο τροπολογίες στην Πολιτική Επιτροπή για να αναφέρω περισσότερο τις απόψεις του Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενέργεια. Τέλος, πρέπει μέσα σε αυτή τη θητεία και σύντομα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ΕΠΕΞ με την αντιπροσωπεία της οποίας προείδρευα να σχολιάσει περισσότερο το Μάρτιο ίσως και να κάνει προτάσεις για τροπολογίες στην αυτή στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ. Επίσης προτάθηκε να γίνει μια δεύτερη έκθεση Βατάνεν για τις σχέσεις με τον ΝΑΤΟ αφού υπάρχει αυτή η νέα στρατηγική αντίληψη και εμείς ασχολούμαστε περισσότερο στο μέλλον με θέματα άμυνας και στρατηγικής, θα έπρεπε να το ξανασυζητήσουμε και να πάρουμε μια θέση. Αυτά. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό το τελευταίο μέρος θα σας έλεγα ότι πράγματι ήρθαμε σε επαφή με την ομάδα της Μαγδαληνής Ολμπράιτ και θα είναι η ομάδα αυτή στις Βρυξέλλες το μήνα αυτόν, αλλά δυστυχώς όταν εμείς θα είμαστε στο Στρασβούργο δεν μπορούμε να συναντηθούμε λοιπόν. Θα ζητήσουμε νέα συνάντηση κατά τον Ιανουάριο για να έρθει να μας πει τι εργασίες εκτελεί τελευταία. Επίσης στον Όρφολκ των Ηνωμένων Πολιτειών θα συναντήσουμε τους στρατιωτικούς και θα οργανώσουμε κάποια ή ακρόαση ή έκθεση για το θέμα των σχέσεων με τον ΝΑΤΟ. Παραμένει σημαντικό για μας, το βλέπετε. Έχουν ζητήσει πολύ το λόγο. Η κυρία Λούζινγκ πρώτα. Η πρώτη μου ερώτηση αναφέρεται σε αυτό το οποίο ανέφερε τελευταίο ο πρόεδρος. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει αυτό το, αυτή τη διαδικασία εμπλοκής του Κοινοβουλίου ή της υποεπιτροπής στο στρατηγικό προγραμματισμό του, του ΝΑΤΟ είναι κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι διότι είπατε ότι θα θέλαμε να συζητήσουμε αυτό ή εκείνο εγώ θα ήθελα να έχω τη δικιά σας αξιολόγηση είναι δυνατόν με τις ενδιάμεσες ε, εκθέσεις ε, που έχουμε ε, για την μεσοπρόθεσμη στρατηγική του ΝΑΤΟ μπορούμε να διαμορφώσουμε ιδέα και να εμπλακούμε στη διαδικασία είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα ήθελα να μου εξηγήσετε διότι αντιλαμβάνουμε ότι η στρατηγική συζήτηση έχει ολοκληρωθεί και προσπαθούμε να συμμετάσχουμε και να εμπλακούμε εμπλακούμε και σε αυτή την πτυχή. Πώς λοιπόν ε, μπορούν να εμπλακούν ε, τα δικά μας θεσμικά όργανα στη συζήτηση αυτή. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται ε, σε ένα ψήφισμα το οποίο έχει συμφωνηθεί το 370. 6 σχετικά με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Διότι αν συζητάμε για το Αφγανιστάν είναι βασικό να έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το τι διαδραματίζεται εκεί. Και από το ψήφισμα αυτό βλέπω ότι καταδικάζουμε την, ε, ε, την στάση των ε, των ε, ε, Αφγανών οι οποίοι συλλαμβάνουν και κρατούν ομίλους και μετά ο Ρόμπερ Πέικ είχε πει ότι ουσιαστικά να το κοιτάζει να προστατεύσει τους ε, ή να επιτεθεί κατά ε, στρατιωτικών στόχων. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω πώς ε, συνδέεται αυτό με το ψήφισμα το οποίο προαναφέραμε και ιδίως όσον αφορά τα διάφορα στοιχεία. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ. Ήταν η πρώτη μου επίσκεψη και μου συνεδρίαση του ΝΑΤΟ ήταν ε, περίεργη εμπειρία. Δεν έχουμε και πολύ καλή φήμη, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχα έτσι κάπως εχθρική υποδοχή από τους Βρετανούς ε, ε, βουλευτές. Δεν γνώριζα αυτή την έκθεση. Η κοινοβουλευτική συνέλευση δεν έχει επίσημο ρόλο στο ΝΑΤΟ. το οποίο μία συνθήκη είχε αντίθετα από την Ένωση, που χρονολογείται από το 1948. Δεν χρειάστηκε να κάνει καμιά ε, μεταρρύθμιση, παρόλο που έχει ενσωματώσει στο θεματολόγιο του θέματα τα οποία παλαιότερα ούτε καν μπορούσαμε να φανταστούμε, όπως τρομοκρατία, κλιματική αλλαγή, ε, κυβερνοασφάλεια κτλ. κτλ. κτλ. Ε, με ανησυχεί λοιπόν, με ανησυχεί επικάλυψη των εργασιών μεταξύ Βρυξελών και ΝΑΤΟ ε, εις ό,τι αφορά και τον στρατηγικό σχεδιασμό και την σχετική επιτροπή. Ήταν κάπως λοιπόν σουρεαλιστική η εμπειρία, ενδιαφέρουσα όμως. Ε, και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι και μια έκθεση, δεν θυμάμαι το όνομα, ενός Νορβηγού νομίζω κυρίου, για το θέμα ε, της στρατηγικής αναθεώρησης του ΝΑΤΟ και των στρατηγικών αποστολών ε, που τώρα θα ονομάζεται Ατλαντικό Συμβούλιο και υπήρχε μόνο μία παράγραφος για τις σχέσεις μεταξύ ε, Ένωσης και ΝΑΤΟ και η συνθήκη της Λισαβόνας δεν αναφερόταν πουθενά να προσθέσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφερόταν ως μια διεθνή οργάνωση όπως τα Ηνωμένα Έθνη, κάπως έτσι. Δηλαδή όλα αυτά τα λέω για να καταλάβουμε την οτροπία του ΝΑΤΟ και των βουλευτών που είναι εθισμένοι στο ΝΑΤΟ και μας υποτιμούν εδώ εμάς ε, από την άλλη μεριά δηλαδή στις Βρυξέλλες που είμαστε και εμείς στην ίδια πόλη αλλά από την άλλη μεριά όπως έλεγε η κυρία εκδεξιών ζητώ συγγνώμη γιατί δεν συνεκράτησα το όνομά της εντύπωση η μου έκανε ότι και για την Αταλάντη υπάρχει μια αντίστοιχη εντελώς παράλληλη και εντελώς ανεξάρτητη από τη δική μας επιχείρηση. Όπως αυτό που κάνουμε εμείς με την Αταλάντη, ακριβώς το ίδιο κάνει και το ΝΑΤΟ. Ε, δεν χρειάζεται λίγο καλύτερο συντονισμός. Ερωτώ. Ο κύριος Καλτιέρη, ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να συμφωνήσω με τον Πρόεδρο Σερουσφόρσκι που είπε ότι χρειάζεται εντονότερος και εντατικότερος διάλογος. με τον ΝΑΤΟ που έχει ξεκινήσει μια σχετική διαδικασία ανοιχτή σε εξωτερικές συνεισφορές και που νομίζω ότι άπτεται ζωτικών θεμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού του Κοινοβουλίου, το ρόλο του στην συμμετοχή της προσπαθίας ορισμού της CSDP, όπως τη λέμε πλέον τη σήμερα ημέρα. Και όχι SDP μόνο. Όχι. Και υπάρχουν διστάμενες, τέλος πάντων διαφορετικές υπόψεις, άποψεις, ε, μια πιο παραδοσιακή, έτσι ενδεχομένως κάπως πιο παλαιά σχολής, για να μην πω απειρχιωμένη, και συγχρόνως μια, άποψη που θέλει να οθήσει τον ΝΑΤΟ όχι μόνο να αντιμετωπίσει την εσωτερική ασφάλεια, αλλά να αντιμετωπίσει και εξωτερικές, εκτός δηλαδή των γεωγραφικών του ορίων κρίσης. Και γι' αυτό ο συντονισμός είναι πολύ σημαντικός. Και πολύ σημαντική είναι και η συμμετοχή μας στην διαδικασία αυτή της ε, σχεδιακής, ε, του σχεδιακού προγραμματισμού, σχεδιασμού. Είναι δική μας απόφαση, όπως είπε και ο πρόεδρος Ντονζό, μέσω της ε, πρόσκλησης στην κυρία Ολμπράιτ, να αναπτύξουμε αυτό το ρόλο περαιτέρω. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της συμπληρωματικότητας και θα ήταν ενδιαφέρον στα πλαίσια αυτά να αξιολογήσουμε ε, την συμπληρωματικότητα και να τη συγκρίνουμε πόσο την ε, αξιολογεί το ΝΑΤΟ και πώς ε, η ΕΟΑ διότι θα ήθελα να ξέρω εάν μπορεί να συμφωνήσει η πλευρά του ΝΑΤΟ και ε, η ε, πλευρά της Ευρώπης για το που υπάρχει επικάλυψη και που όχι. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια καλή και ε, ορθολογιστική βάση για μελλοντική συζήτηση. Δεύτερον, έχω δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Ζάριους Βόσκη. Καταρχήν, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές συζητήσεις γενικώ. Και αν ναι, πώς μπορεί να έπαιξε ρόλο η πρόταση του Μετβέντεφ. Και θέλω να επανέλθω και στο θέμα του Αφγανιστάν. διότι ο πρόεδρος ε, ε, Ομπάμα σήμερα παρουσιάζει τις νέες ιδέες του. Ήδη τη Δευτέρα διαβάσαμε στις εφημερίδες ότι μαζί με, ε, με Ευρωπαίους ηγέτες ε, στους οποίους τηλεφώνησε ε, προσπαθεί να ε, αναβιώσει την προσπάθεια στο Αφγανιστάν αλλά πολλοί δεν συμφώνησαν μαζί τους ε, ε, στην Ευρώπη και ιδίως ο κύριος Σαρκοζή. Είπατε ε, υπήρχε μεγάλη διαφορά απόψεων από έναν Γεωργιανό που ζητούσε μεγαλύτερη επέμβαση και του άλλους οι οποίοι ζητούσαν πλήρη απόσυρση. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται. Ε, στο ΝΑΤΟ η πλειοψηφία είναι αρνητική, είναι ε, σκεπτική σχετικά με μία εμπλοκή στο Αφγανιστάν ή πώς γενικώ θα μπορούσαμε να έχουμε ερμηνεύσει αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. το, έκανα... το θέμα του τι έγινε στο Εδιμβούργο μας ενθαρρύνει να αρχίσουμε τώρα καινούργιε συζητήσει που μπορεί να απαιτήσουν να τρει ώρε. Εγώ ήθελα απλώ να αναφέρω ποιο ήταν το γενικότερο κλίμα. Σας είπα, ζήτησα από την ΕΠΕΞ να ασχοληθεί με το θέμα των σχέσεών μας με το ΝΑΤΟ, γιατί μέχρι τώρα είναι, δεν είναι ικανοποιητικέ. Είναι όλα διαφορετικά, δεν υπάρχει καμία συνεννόηση, όλα αλλιώτικα. Εμείς έχουμε το Κόρτενμπεργκ, εκείνοι έχουν άλλες εγκαταστάσεις, όλα διαφορετικά και διαφορετική νοοτροπία. Από τα ίδια εθνικά κοινοβούλια αυτοί που πάνε στο ΝΑΤΟ και αυτοί που πάνε σε, μας συναντάνε εμάς άλλα λένε. Μιλάνε άλλη γλώσσα. Και αυτά που είπε ο κ. Στάνο όλα ισχύουν. Συχνά στο Εδιμβούργο η συζήτηση έδειχνε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική για το ΝΑΤΟ, ευρωπαϊκή άποψη σαν να υπήρχε κάποια περιφρόνηση προς την Ένωση, να έλεγαν «Α, τι είναι η Ένωση, δεν είναι τίποτα, εμείς έχουμε την εξουσία και τα μέσα». Άρα χρειάζεται περισσότερος διάλογος. Γιατί και εμείς αργά αλλά σταθερά θέλουμε περισσότερο στρατηγικό ρόλο, εγώ το αποκαλώ νατοποίηση της Ένωσης, δηλαδή περισσότερες δικαιοδοσίες για hard security και όχι μόνο soft. Το ιδεώδες θα ήταν να εξευρωπαϊστεί το ΝΑΤΟ βέβαια, ιδίω μετά την επιστροφή της Γαλλίας σε αυτό. Γιατί το ΝΑΤΟ δεν αφορά μόνο τεθωρακισμένα και στρατιώτες, έχει και πολιτικές αποστολές για θέματα δικαιοσύνης και άλλα. και ως τα οποία θα μπορούσε να συμβάλλει και η Ένωση όπως το Αφγανιστάν που είναι πολύ μικρός ο ρόλος της. Πρώτο ερώτημα λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε και εμείς. Εμείς είμαστε παρατηρητές, δεν ψηφίζουμε για τα ψηφίσματα αυτά, είμαστε παρατηρητές και παρατηρήτριες. Δεν είμαστε βέβαια απλώς προσκεκλημένοι, αλλά υπάρχουν και οι Νεοζηλανδοί και οι Ιρανοί. Εμείς έχουμε το δεύτερο υψηλότερο καθεστώς δηλαδή. Μπορούμε να συμμετέχουμε, να προτείνουμε, να μιλούμε, απλώς δεν μπορούμε να ψηφίζουμε. Άρα είμαστε σε θέση να εκφράσουμε τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα ασφαλείας και άμυνας προς την Κοινοβουλευτική Συνέλευση που όπως είπε και ο κύριος Τάνοκ δεν έχει πολλές δικαιοδοσίες, δεν βασίζεται σε καμία συνθήκη αλλά καθορίζει και αυτό κάπως την πολιτική του ΝΑΤΟ και πρέπει τα ψηφίσματά του να τα λαμβάνουν υπόψη οι στρατιωτικοί Αν μπορούμε λοιπόν, αφού μας καλούν, να συμβάλλουμε και εμείς κάπως στη συγγραφή των εγγράφων τους, τότε θα έχουμε παίξει κάποιο ρόλο. Αυτή είναι η απάντησή μου στο πώς θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε. Δεν θα απαντήσω για το Αφγανιστάν την ερώτηση, γιατί δεν έχω τις γνώσεις που απαιτούνται, ούτε και το χρόνο αν είχα τις γνώσεις. Δύο ερωτήσεις έθεσε. Ο συνάδελφος, να εδώ δεν το βλέπω. Μετβέντεφ. Α, όχι, την πρόταση του Μετβέντεφ. Για ποια πρόταση του Μετβέντεφ, για τη νέα αυτή δομή. εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, δεν μπορώ να σου πω τι σκέφτεται με την Όχι, δεν είναι δικέ μου θέσει αυτά, δεν με αφορούν αυτά. Και στην προηγούμενη θητεία στην ΕΠΕΞ είχαμε πει να δείξουμε φρόνηση ως προς αυτήν την νέα προσέγγιση του Μετβέντεφ που έχει σκοπό να αποδυναμώσει τις δομές της Δύσεως και της Κέπας δεν είναι έντιμη προσπάθεια και είναι πονή. Μα εγώ το ρώτησα πολύ αθώα. Θα το σκεφτεί. Όχι. Όχι. Είτε συμφωνείτε είτε όχι. Εμείς και συζητάμε μόνο σοβαρά θέματα και όχι πολιτικές μπλόφες. Τώρα για τον Ομπάμα. Απ' τη μία μας κάλεσαν οι Βρετανοί με τον Ράσμουσεν που ζήτησαν μεγαλύτερο μερίδιο των Ευρωπαίων στα βάρη του ΝΑΤΟ. Ε, κάτι ανάλογο είπε και ο Ομπάμα, αλλά υπήρξαν πολλών ειδών αντιδράσεις, από σιωπή μέχρι απόσυρση, μέχρι περιορισμένης εντολής αποστολή στρατευμάτων, α, όλα τα είπανε. Έτσι κάνουν οι Αμερικάνοι. Ε, όλα. Δεν είναι θέμα καθαρά του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, άρα δεν υπάρχει αυτόματη υποχρέωση να συμβάλλουμε, αλλά Μερικοί λένε ότι θα είναι μια δοκιμή των δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ. Μάλλον σωστό είναι αυτό. Μια αποτυχία θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία του ΝΑΤΟ. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια εξαρτάται από το ΝΑΤΟ για την πυρηνική αποτροπή τουλάχιστον και μπορεί να συμπληρωθεί από, τη δική, από τις δικές μας αμυντικές δυνατότητες όσο λίγες και να είναι προς το παρόν. συμπληρωματικότητα και είπες. Προτιμώ να εργαζόμαστε συμπληρωματικά παρά με βάση τις υποχρεώσεις που ανέφερε ο κύριος Τάνοκ. Ο διπλασιασμός των Αμερικανικών δυνάμεων δεν νομίζω ότι θα τύχει διαχείριση από το ίδιο στρατηγείο. Ναι, λοιπόν, συμπληρωματικότητα είναι κάτι που μπορούμε εμείς να εφαρμόσουμε. Περισσότερες επαφές μεταξύ ΝΑΤΟ και Ένωσης, αλλά με βάση εμάς, εμάς. εμάς. Και εγώ θα πήγαινα κανονικά σε αυτή την αντιπροσωπή, αλλά είχαν λυμμένες υποχρεώσεις. Το συνέδριο του κόμματό μου δεν μπόρεσα να πάω στο Εδιμβούργο. Ήθελα όμω ήθελα. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην προηγούμενη θητεία είχα τονίσει επανειλημμένος ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν το είπα αυτό γελάσανε όλοι. Αλλά εγώ το είχα διαπιστώσει και με τα μάτια μου σε μια προηγούμενη ζωή όπως λένε. Και τώρα το διαπίστωσαν κι άλλοι συνάδελφοι και κατάλαβαν ότι είναι κάτι το πραγματικό αυτό που είχα πει. Το άκρο όταν είναι ότι πρόκειται για τα ίδια στρατεύματα οι ίδιοι στρατιώτες είναι. Δεν υπάρχει για καμία χώρα άλλη δύναμη ευρωπαϊκή και άλλη για το ΝΑΤΟ. Τους ίδιους θέλουν, τους ίδιους με διαφορετική επομίδα ή διαφορετικό μπερέ. Αλλά οι ίδιοι είναι και οι ίδιες. Πρέπει λοιπόν αυτό να ξεκαθαριστεί ως το δυνατόν συντομότερα. Η φύση των δύο οργάνων φυσικά είναι διαφορετική. Δεν χρειάζεται καν να το πούμε πόσο διαφορετική είναι. Υπάρχει όμως ανταγωνισμός. Θυμηθείτε τα battle groups και τη rapid intervention force. Οι μεν έκαναν το ένα, οι δε το άλλο. Ενώ πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Υπάρχει κίνδυνος επικάλυψης και των στρατηγίων και των σχεδίων. Απολύτως. Διότι υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτό πρέπει να το δούμε κατάματα και δεν χρειάζεται κανένα νόημα να το παραβλέπουμε. Πρέπει να μειωθεί ο ανταγωνισμός αυτός, γιατί δεν εξυπηρετεί τίποτε. Λοιπόν, είναι τεράστια η προβληματική που τίθεται εδώ και ελπίζω κάποια μέρα να τη συζητήσουμε γιατί αξίζει τον κόπο είναι μια πραγματικότητα. Οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ένωσης ποτέ δεν ήταν απλές βέβαια. Θυμάμαι την περίοδο κατά την οποία ο κύριος Σολάνα που ήταν τότε ακόμη γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ μπορούσε να έρθει να πιει έναν καφέ στα ανεπίσημα γεύματα των υπουργών. Μπορούσε να έρθει για καφέ, το ξαναλέω. Ξέρετε τι εννοώ. Από τότε άλλαξαν τα πράγματα και πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη πριν μπορέσουμε να πούμε ότι τα δύο όργανα συμπεριφέρονται το ένα προς το άλλο ενηλίκως. Γιατί πρόκειται για θέμα ασφάλειας και των στρατιωτών και γενικότερα. Ευχαριστούμε. κυρία Λούζινγκ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό σαν βουλευτές πρέπει να προσπαθήσουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς αυτή τη διαδικασία διότι στις τελευταίες συνεδριάσεις εδώ έχουμε μιλήσει για συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και έχω όλο και περισσότερο την εντύπωση ότι όλο και περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη ε, ζητούν ε, περισσότερο ε, περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευκολύνουν το ΝΑΤΟ και να το αποσυμφορήσουν. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή ε, είναι μία συμπληρωματική διεργασία αλλά βλέπω ότι ε, μετατίθεται η λήψη των αποφάσεων όλο και περισσότερο προς το ΝΑΤΟ. Αν δω ας πούμε τους στρατηγικούς στόχους την ε, κατάργηση των, ε, ε, των εθνικών προκαταλήψεων, το caveat που λένε διότι οι Γερμανοί θα έπρεπε να αποφασίσουν μόνοι τους εάν θέλουν να επέμβουν στο Νότιο Αφγανιστάν ή όχι. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και μπορεί κανείς ε, να, να χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους. Παραδείγματο χάρη ε, οι αρχές αυτές θα καταργηθούν με την εξέλιξη του ΝΑΤΟ και άλλα πολλά όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο συνολό της ίσως, αλλά τα κράτη-μέλη πρέπει όλο και περισσότερο να εμπλέκονται, όλο και περισσότερο να πληρώνουν και έχουν όλο και λιγότερη τη δυνατότητα να συναποφασίσουν για μία ενέργεια. Και αυτό με εκπλήσει πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπω ότι ε, υπάρχουν ελάχιστη ελάχιστα μέλη αυτής της αντιπροσωπείας που ενδιαφέρονται για αυτή τη συζήτηση, πράγμα το οποίο μας δείχνει ε, ποια είναι η δυνητική σημασία των αλλαγών του ΝΑΤΟ για μας. Επίσης, όσον αφορά την ε, αμυντική και διάρθρωση ή τη διάρθρωση ασφαλείας. Υπάρχουν συζητήσεις και εγώ θα πρότεινα ή στην ε, Υποεπιτροπή Ασφαλείας να ασχοληθούμε και εμείς με αυτό το οικοδόμημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος όλα αυτά τα ερωτήματα αποδεικνύουν ότι χρειάζεται συζήτηση με περισσότερους από τρεις ευρωβουλευτές στην αίθουσα. ή πέντε τέλο πάντων ευρωβουλευτέ εντό τη αίθουσα. Σχήμα λόγου είναι, καταλάβατε τι εννοώ. Λίγοι θέλω να πω. Λίγοι. Ε, Πάντω ε, νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να έχουμε μια συζήτηση επί δύο ώρες με έναν εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ για να συζητήσουμε την έκθεση Βατάνεν και άλλα. Όντως, υπάρχει πρόβλημα με τον ανταγωνισμό με τον ΝΑΤΟ. Είναι χαρτοφυλάκιο που πρέπει να πάρει η καλό πράγμα αρκεί να είναι θεμητός έτσι επιτάσει η ελεύθερη αγορά. Να ακούσουμε και το Μισελ Μπαρνιέ τι έχει να πει. Τέλος πάντων, αστείευομαι. αστείευομαι. Είναι σοβαρό το ζήτημα. Και ήθελα να πω ότι δεν αντιμετωπίζεται έτσι στο γόνατο. Εντάξει, όχι στο γόνατο, αλλά τέλο πάντων ε, εν παρόδο και με τόσο μικρή παρουσία ευρωβουλευτών. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου είμαστε μαζί με το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ, το Αφγανιστάν. Το, με το ΝΑΤΟ εννοώ το Κόσοβο και το Αφγανιστάν. Τέλο πάντων, δεν μπαίνω σε περισσότερε λεπτομέρειε. Μπορούμε να το συζητήσουμε και με τον κύριο Αλμπερτίνη. Πάντω ο πρόεδρο και ο υποφαινόμενο πιστεύουν ότι χρειάζεται σε μεγαλύτερο βάθο συζήτηση για το θέμα. Σχέσει Ε ΝΑΤΟ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ναι, εν κατακλείδη πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με την ΑΦΕΤ. Όχι το Δεκέμβριο βέβαια, γιατί τεχνικά δεν είναι δυνατόν να είμαστε παρόντες, αλλά ε, τον Ιανουάριο που θα έρθει η Μαντλινόρ Μπλάιτ να έχουμε τη δυνατότητα να οργανώσουμε έτσι μια πιο ουσιαστική συνάντηση. Για το θέμα του ανταγωνισμού μεταξύ ημών και του ΝΑΤΟ ή της παραπληρωματικότητος, ναι, συμφωνώ και επιχειρησιακά. Είδαμε τις 22 επιχειρήσεις που έχει αναλάβει η Ένωση. Το Αφγανιστάν είναι μια κρίσιμη βεβαίως περίπτωση. Η Σομαλία επίσης, αλλά η Αταλάντη για τη Σομαλία δεν οδήγησε σε ανταγωνισμό γιατί το ΝΑΤΟ έχει πολύ λίγα ε, στρατεύματα σε σχέση με την Ένωση και ε, νομίζω ότι οι περισσότερες περιπτώσεις επί των οποίων οι επιχειρήσεις της PSD ήταν επιτυχής ήταν ε, παραδείγματα όπου δεν υπήρχε ανταγωνισμός αλλά συμπληρωματικότητα με τον ΝΑΤΟ. Βλέπε Κόσοβο η Γεωργία. Η Γεωργία δε είναι αποκλειστικότητά μας, έτσι. Αλλά πάντως τα προβλήματα που θέσατε είναι πραγματικά κάπως ε, λιγότερο έτσι, φανερά σε σχέση με τις επιχειρήσεις, αλλά υπάρχει αυτό και θα επανέλθουμε από τις αρχές του 2010 και μετά, γιατί είναι θέμα ε, που μπορούμε να εμβαθύνουμε. Και θα το συζητήσουμε και με την κυρία Άστον. Πώς μπορούμε με την ε, νέα συνθήκη, με την νέα αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής ε, Οργάνωσης να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τον ΝΑΤΟ. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο, αύριο το πρωί στις 10 η κυρία Άστον θα υπάγει στην ΑΦΕΤ. Στο ημικύκλιο. Στο ημικύκλιο. Και εμείς θα τα ξαναπούμε στις 10 Δεκεμβρίου. Και συμφωνώ πλήρως με την κυρία Λούζινγκ για την ε, μικρή συμμετοχή στη συζήτηση Πρέπει να πείσουμε τους αδέρφους να ενδιαφερθούν περισσότερο.